αναφορών. Εγώ λέγομαι Ρομπέρτο Γιόντα, γι' αυτό δεν ε, μίλησα. Νομίζαμε ότι ο Ρενάτο Λέλη ήταν αυτός ο οποίος θα μιλούσε. Εσείς, για ποια αναφορά είστε. Για την 57 του 2018, δεν ξέρω αν είναι αυτή η δική μου που είναι αυτή που έχετε υποβάλει με 100 υπογραφές. Οι κύριοι που σας συνοδεύουν είναι αναφέροντες από άλλες αναφορές. Όχι, όχι, είναι με τη δική μου την αναφορά. Ωραία, θα κάνουμε το εξής. Έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ. Καταρχά, ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του παρισταμένου και όλου εκείνου που ε, δίνουν αυτή τη μάχη ε, πολιτισμού. Λυπάμαι που το λέω, είναι μια μάχη δυστυχώς που πρέπει να προχωρήσει διότι είναι απαραίτητο να αποφύγουμε την τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Στην Ιταλία είναι υπερβολικό ο εμβολιασμό και ε, γίνεται διάκριση ε, των Ιταλών παιδιών ενώπιον των υπόλοιπων Ευρωπαίων διότι προβλέπεται και ε, ότι για την περίοδο 0 έως 6 ετών τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο αν δεν έχουν εμβολιαστεί και θεωρούμε ότι αυτή είναι διάκριση σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά ε, στις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν... Ε, ε ε, μπορεί ένα παιδί να φοιτήσει στο σχολείο ε, στα έξι έτη αν δεν έχει ε, εμβολιαστεί. Έχω εδώ μια έκθεση του δόκτωρα Φράγκη που φαίνεται προφανώς ότι μεταξύ αυτών των εμβολίων υπάρχουν διάφορα εμβόλια όπως για παράδειγμα το MPR που περιλαμβάνουν αλουμίνιο και άλλα μέταλλα τα οποία είναι τοξικά. Γι' αυτό εγώ λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει θέση και να τοποθετηθεί γιατί βάσει του άρθρου 6 τη Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση η δημόσια υγεία είναι μία από τι προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να ε, αποτανθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μία πιθανή πρόταση που θα μπορέσει να εγγυηθεί την ασφάλεια και την υγεία όλων των Ιταλών υπηκών που δυστυχώ υποβάλλονται από παιδική ηλικία σε αυτά τα 10 εμβόλια. Εγώ επίσης θεωρώ ότι εδώ ολοκληρώνω την παρέμβασή μου και ε, ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα αναλάβει ευθύνες, διότι η υγεία των παιδιών είναι η υγεία του μέλλοντός μας. Και ελπίζω να θεωρηθεί ε, εξίσου σημαντική αυτή η μάχη για το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η υγεία υπερπάντων. Ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κυρία Ίγκον Βέρσεν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο νόμος που εγκρίθηκε στην Ιταλία και κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των παιδιών μέχρι τα 16 έτη, ώστε να έχουν πρόσβαση στο σχολείο είναι ένα θέμα. Επίσης, ε, πρόσφατα είχαμε ένα θέμα που προέκυψε κάπως επίγον ε, το θέμα της ηλαράς ε, που μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από τα εμβόλια. Υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό. Ο Ιταλικός νόμος έχει οδηγήσει σε μία συζήτηση στην Ιταλία και στην ουσία η σημερινή αναφορά είναι μια συνεισφορά σε αυτή την ίδια συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πολλά περιθώρια χειρισμών σε αυτό το θέμα, γιατί τα ζητήματα υγείας και πρόνοιας ε, είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτά πρέπει να θεσπίζουν τα προγράμματα εμβολιασμού. Όπως και να έχει όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη-μέλη ε, στην προσπάθειά τους να καλύψουν τον πληθυσμό ε, με εμβολιασμό έναντι ασθενειών που μπορούν να αντιμετωπιστούν με εμβόλια. Ε, θέλουμε να έχουμε υψηλό ποσοστό εμβολιασμών για να διαφυλάσσουμε τη δημόσια υγεία. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες για τους εμβολιασμούς με σκοπό την ε, υγεία και την ασφάλεια. Υποστηρίζουμε τον εμβολιασμού. Οι Υπουργοί Υγεία επίση της Ευρωπαϊκή Ένωσης έχουν υιοθετήσει μία θέση ε, σύμφωνα με την οποία ταυτοποιούνται οι ασθένειε που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον εμβολιασμό και αναφέρεται η δράση που μπορεί να ληφθεί εναντίον του. Επίση, προωθείται η πληροφόρηση για τι συγκεκριμένε ασθένειες γιατί θέλουμε το κοινό να γνωρίζει τις πληροφορίες αυτές και να γίνεται ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Επίσης, ε, το Σεπτέμβρη ε, θα γίνει μια παγκόσμια διάσκεψη για τον εμβολιασμό σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ε, για το 2050 του 2019 να πω ότι έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες που αφορούν στους εμβολιασμούς και υπάρχουν σοβαροί έλεγχοι που γίνονται προτού δοθεί οποιοδήποτε εμβόλιο στην κυκλοφορία. Ευχαριστώ. πολύ. Και τώρα περνάμε στους ευρωβουλευτές. Ε, υπάρχει κάποιος ο οποίος ε, θα ήθελε το λόγο. Η κυρία Κυρτον Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον αναφέροντα που ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η αναφορά τονίζει μια πολύ ανησυχητική τάση που έχει αναδυθεί στην Ευρώπη. Έχουμε επιστροφή στα κράτη-μέλη ασθενειών που στο παρελθόν θεωρούσαμε ότι είχαν εξαλειφθεί αποτελεσματικά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, τον Αύγουστο, είχαμε 230 περιστατικά ηλαράς. Οπότε χάσαμε το καθεστώς ε, της χώρας που έχει απαλλαγή από την ηλαρά στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συζήτηση για τον εμβολιασμό ήταν εδώ και χρόνια μια πολύ ζωντανή συζήτηση. Σύμφωνα με τις ε, ιατρικές ε, έρευνες, Ε, υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία τα οποία ε, στην αρχή φαινόταν αξιόπιστα, μετά καταφέραμε να δείξουμε ότι είναι παραπληροφόρηση και υπήρξαν και γιατροί οι οποίοι διαγράφηκαν από τους καταλόγους ακριβώς επειδή διέδιδαν αυτή την παραπληροφόρηση. Κάποιες ασθένειες δεν πρέπει πλέον να εμφανίζονται στις ε, προηγμένες χώρες μας. Είναι μεγάλο το πρόβλημα γιατί τα fake news και η παραπληροφόρηση είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα γι' αυτό, ε, για το πώς δηλαδή εγκρίνονται τα φάρμακα. Υπάρχει παραπληροφόρηση που παίζει με τους φόβους των γονιών μικρών παιδιών. υπάρχει αυτή, αυτός ο υπενιγμός ότι το παιδί κινδυνεύει αν εμβολιαστεί και κανένας γονέας δεν θέλει να θέσει το παιδί του στο κίνδυνο. Εμείς ως δημόσιες υπηρεσίες, ως πολιτικοί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση. Λυπάμαι που είμαι έτσι αυστηρή και λίγο ξερή, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να πούμε ανοιχτά και στην Επιτροπή Αναφορών όταν έρχονται αναφορές που θέτουν τέτοια ζητήματα, που γύρουν τέτοιες ανησυχίες. Ένα από τα προβλήματα που εγώ προσωπικά έχω με αυτές τις τάσεις που είδαμε σε μια σειρά χωρών, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και αλλού στον κόσμο, επίσης στις Ηνωμένε Πολιτείε, είναι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των fake news για την διάδοση μύθων, για τη διάδοση τρομακτικών ιστοριών για τον εμβολιασμό που τελικά οδηγούν σε μείωση της κάλυψης του πληθυσμού μας ε, έναντι ασθενειών που θα πρέπει ήδη να έχουμε ξεχάσει ε, και οι οποίες είναι ε, απειλητικές για την υγεία, για τη ζωή, συγγνώμη τα κράτη-μέλη έχουν συγκεκριμένες πολιτικές υγείας ε, και τις γνωρίζουν. Δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς να θέτει υπό αμφισβήτηση τα αυστηρά κριτήρια που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Εντάξει, πάντα πρέπει να αμφισβητούμε και να διαρωτόμαστε, όμως πρέπει να πούμε και ξεκάθαρα ότι στην Ευρώπη για να μπορούμε να βγάλουμε ένα φαρμακευτικό προϊόν στην αγορά, το οποίο προορίζεται για εμβολιασμού, πρέπει να έχουμε κάνει συγκεκριμένε αναλύσει, να έχουμε τηρήσει συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλεία. Άρα, συστήνω αυτές οι αναφορές να πάνε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας όπου εκεί αντιμετωπίζονται τα ζητήματα αυτά με βάση το περιεχόμενο και τους κανονισμούς για τα φάρμακα. Δεν βλέπω να μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς ως κοινοβούλιο βάσει των όσων έχουν κατατεθεί εδώ στην Επιτροπή Αναφορών και θα ήταν μεγάλος κίνδυνος να συνεχίσουμε να ταΐζουμε με υποστήριξη και πληροφορίες μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που τρέχει σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να πω ότι ε, και εγώ συμφωνώ ότι είναι επικίνδυνο να παντίζουμε σε αυτά τα νερά. Στον εμβολιασμό ε, υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες ε, σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις όμως το σημαντικό είναι ότι για τους ανθρώπους τα καλά είναι μεγαλύτερα. Το συμπέρασμα της συναδέλφου μπορώ να πω ότι είναι σωστό. Αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε την εσωτερική αγορά, έχουμε συγκεκριμένες άδειες για τα φάρμακα και χρειαζόμαστε και μια στρατηγική γιατί ε, όταν στη μία χώρα γίνεται κάτι σχετικά με τους εμβολιασμού και από την άλλη στη διπλανή χώρα υπάρχει διαφορετική στρατηγική, δεν είναι ωραία η εικόνα. Ε, καλό είναι να μην υπάρχει αυτό έτσι. Γι' αυτό καλό θα ήταν να στείλουμε αυτή την ε, ε, αναφορά προς περαιτέρω εξέταση για να μπορούν τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν ναι μια πιο σαφή στρατηγική και η εναρμόνιση θα βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ουσιώδους σημασίας. Ε, θα σας δώσω δύο λεπτά ε, στον αναφέροντα, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος ε, θέλει το λόγο από την Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι στην τεκμηρίωση που σας έχω ε, στείλει υπάρχουν τα στοιχεία της IFAR. Η IFA είναι ο Οργανισμός Φαρμάκων, ο ΕΟΦ ο αντίστοιχος και εδώ πρόκειται στοιχεία. Δεν πρόκειται για κάποιο τρελό γιατρό ο οποίος γνωμοδοτεί στην κλινική του στον Άρη, αλλά ο Οργανισμός Φαρμάκων αναφέρει 31 ε, ε, περιπτώσεις σε 100.000 αντενδείξεων. Ε, νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή, γιατί άκουσα από του ε, βουλευτές που μίλησαν πριν από εμά ότι πρόκειται για fake news, για ψευδεί ειδήσει. Νομίζω ότι κάθε φορά που πρόκειται για παιδιά πρέπει να σκεφτούμε 10, αν όχι και 10.000 φορέ περισσότερο για το τι μπορούμε να κάνουμε για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των παιδιών που βρίσκονται σε πολύ ευαίσθητη ηλικία. Εγώ ελπίζω λοιπόν το Κοινοβούλιο να μπορέσει τουλάχιστον όσον αφορά την ασφάλεια των ε, εμβολίων να κάνει κάτι περισσότερο από όσα έχει γίνει σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι που μου δώσατε το λόγο. Perfecto. Τέλεια. Μετά από τα όσα είπαν οι αναφέροντες, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συνάδελφοι της Επιτροπής, η πρόταση της Προεδρίας είναι η εξής να παραπέμψουμε τις αναφορές αυτές ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και Δημόσιας Υγείας, ώστε να μελετήσουν πραγματικά την ουσία του θέματος και εμείς ε, να ολοκληρώσουμε την εξέταση αυτών των αναφορών, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα ακούσαμε και δεδομένου ότι εμείς δεν έχουμε άλλη αρμοδιότητα πέραν αυτού για να συνεχίσουμε να εξετάζουμε τις συγκεκριμένε αναφορές. Συμφωνείτε? Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον ε, Ιταλό αναφέροντα και συνεχίζουμε με την επόμενη αναφορά από κάποιον πολωνικής ηθαγένειας, η οποία φέρει δύο υπογραφές εξ ονόματος της Ένωσης Πράβο ε, Μπέξια σχετικά με την κατασκευή τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων σε περιοχή Natura 2000 στην Πολωνία. Ο αναφέρον είχε διαβιβάσει ότι δεν, μπορέσει, δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Θα δώσουμε λοιπόν απευθείας το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα ε, στον κύριο Ογκίνσκι. Um, Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Οι ανησυχίες μας ε, αφορούν την κατασκευή ενός τερματικού σταθμού εμποροκυματομοτήων στην Πολωνία. Ε, πιστεύουμε ότι θα ε, υπάρχει ε, πρόβλημα στο περιβάλλον αλλά και στην ασφάλεια και ποιότητα της ζωής των, του ντόπιου πληθυσμού. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Επιτροπή, το πρόγραμμα αυτό είναι μόνο στα σχέδια και η υλοποίηση του δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Εάν το πρόγραμμα και ο, η αρχή που θα το υλοποιήσει προχωρήσει σε αυτό, τότε θα πρέπει να ε, καταρτήσει ε, περιβαλλοντική μελέτη, προβλέποντας φυσικά και την ακαιρεότητα του ε, προγράμματος Natura, και επίσης δημόσια διαβούλευση. Ο αναφερόν σε αυτό το στάδιο μπορεί να εκφράσει τις ανησυχίες του. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Νομοθεσία, σε ορισμένες περιπτώσεις τα άτομα μπορούν να αποκτήσουν καθεστώς κόμματος και να συμμετέχουν μάλιστα στις διαδικασίες. Σε αυτό το στάδιο η Επιτροπή δεν, ε, ε, δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίες ευρωπαϊκού νόμου αναφορικά με αυτό το σχέδιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα είναι η σειρά των μελών της Επιτροπής, η κυρία Σδάνοκα. Ε, I hope that the petitioner... Ελπίζω ότι ο αναφέρον βλέπει την συνεδρίαση εφόσον δεν είναι παρόν, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Καταρχάς θα ήθελα να ε, τον ευχαριστήσω για, την, για το ότι έθεσε το, εξέφρασε τις ανησυχίες του τόσο νωρίς. Οι συμπέρασματα της Επιτροπής είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμα παραβιάσεις του νόμου, σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον. Καλό είναι όμως που ε, γνωστοποιείται το ζήτημα. Στη χώρα μου ε, υπάρχουν αντίστοιχα ε, projects, επίσης σε, επίσης σε περιοχές Natura 2000, πάλι με τερματικό σταθμό εμπορικών κυβωτίων. Θα πρότεινα λοιπόν να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά εφόσον υπάρχουν ε, εφόσον υπάρχει πιθανότητα οι αρχές να αποφύγουν την, ε, τη μελέτη περιβαλλοντικού κινδύνου, αντίκτυπου. Νομίζω λοιπόν που, ότι ε, είναι καλό που υπάρχει αυτή η αναφορά και θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να επενθυμίσουν στην Πολωνία ότι πρέπει να εφαρμόζουν και να κινούνται βάσει των ήδη υπαρχόντων κανονισμών. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς, ο Πίτερ ähm, Για τους συναδέλφους να πω ότι τα επιχειρήματα δεν είναι λάθος ε, και θα μπορούσα να συνταχτώ μαζί τους, αλλά και ο αναφέρον έχει δίκιο. Θα ήθελα η Κομισιόν να παρακολουθήσει αυτό το θέμα με την ανάλογη συνέπεια. Είναι ακόμα όταν τα σχέδια αυτά τα μεγάλα είναι στο η φάση του σχεδιασμού, γιατί όταν έχει περάσει αυτή η φάση είναι πιο δύσκολο να διορθωθούν τα λάθη. Καλό είναι λοιπόν με συνέπεια να παρακολουθεί η Κομισιόν αυτά τα σχέδια. Για μένα λοιπόν ε, ε, το θέμα δεν είναι μόνο στρατηγικό, ε, αν θα κρατήσουμε ανοιχτή ή κλειστή την αναφορά. Το θέμα είναι αν μπορούμε να παρακολουθούμε αυτές τις αναφορές, γιατί πολλές φορές τις αφήνουμε ανοιχτές και μετά τις ξεχνάμε. Άρα ίσως καλό θα ήταν για συμβαστική λύση να την αφήσουμε ανοιχτή και να υπάρχει και μια προθεσμία για να μην ξεχαστεί. Γιατί κάποιες φορές ε, έχουμε αυτό το πρόβλημα τη ωραία κοιμωμένη εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. I think we're happy uh, to keep it open. Ε, θα μείνει η ανοιχτή. Ε, νομίζουμε ότι θα υπάρχει περαιτέρω δράση. Ευχαριστούμε. Ωραία, να ολοκληρώσουμε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και θέλουμε να διατηρήσουμε ανοιχτή την εξέταση και να αποστείλουμε επιστολή στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Πολωνίας ε, που θα περιλαμβάνει τα θέματα που θέτει η αναφορά και ε, θα ε, τονίσουμε την ανησυχία των ευρωβουλευτών αυτής της Επιτροπής διότι τον Αύγουστο του 2019 το Πολωνικό Κοινοβούλιο έλαβε απόφαση όσον αφορά τα κοντέινερ σε αυτό το, την περιοχή την οποία πολύ δύσκολα μπορώ να προφέρω της Πολωνίας. Άρα, επειδή ε, υπάρχει και το αίτημα του συντονιστή του ΕΛΚ, ε, όταν θα λάβουμε τις πληροφορίες από τις πολωνικές αρχές, θα γίνει μια δεύτερη εξέταση και ε, στη συνέχεια θα μπορέσουμε να δούμε κατά πόσον θα ολοκληρωθεί το θέμα ή όχι. Προ το παρόν όμω ε, θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δώσει επικαιροποιημένε πληροφορίε για το σχέδιο αυτό, ε, βάσει και των πληροφοριών που σα είπα ότι στι 9 Αυγούστου του 2019 το Πολωνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο ε, και έλαβε απόφαση για αυτό τον τερματικό σταθμό των κοντέινερ. δεν ξέρω αν συμφωνούν οι συντονιστέ. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη αναφορά και να ολοκληρωθεί το θέμα αυτό. Πάμε λοιπόν στην επόμενη αναφορά, επειδή όμως ε, προχωρούμε πολύ γρήγορα, γιατί προβλεπόταν να ξεκινήσει στις 3 και 25 η αναφορά αυτή. Και εδώ έχουμε παρουσία ενός εκ των αναφερόντων, ο κύριος Όλιβερ Στάινερ. Δεν ξέρω αν είστε Όλιβερ Στάινερ. Όχι. είναι ο αναφέρον εδώ της επόμενης αναφοράς, της 2533, δεν είναι εδώ, όχι. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Εδώ η γραμματεία μου λέει ότι σήμερα το πρωί ο κύριος Στάινερ, ο αναφέρον, είπε ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σήμερα το απόγευμα. Επίσης μου λένε ότι έχουμε εδώ τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδια για το θέμα. Επομένως θα συνεχίσουμε με τις αναφορές μας και θα δούμε τι θα κάνουμε. Πρόκειται για την 2553 του 2014 από το Ludwig Μπουλμάιερ, γερμανική σαδαγένεια σχετικά με τα μικροπλαστικά και τα νανοσωματίδια. Μετά, αναφορά 663 του 2015 του Όλιβερ Στάινερ, γερμανικής ηθαγένεια, για τη διαδικασία εγκατάσταση συστήματος καθαρισμού σε όλες τις ευρωπαϊκές μονάδες επεργασίας υδάτων για το φιλτράρισμα των μικροπλαστικών. Κατόπιν, η 783 του 2015 από έναν υπήκο γερμανική ηθαγένεια σχετικά με την απαγόρευση καλλιντικών προϊόντων που περιέχουν μικροπλαστικά. Ε, επίσης, αναφορά 793 του 2015 του Όλιβερ Στάινερ, γερμανικής ηθαγένειας, σχετικά με την απαγόρευση μικροπλαστικών σε καλλιτικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ρουχισμό. Κατόπιν αναφορά 0695, η τελευταία του 2018, και πάλι από κάποιον υπήκο Γερμανία σχετικά με την παρουσία μικροπλαστικών σε βιοστερεά που χρησιμοποιούνται σε γεωργικά λιπάσματα και υλί καθαρισμού λιμάτων. Επειδή ο αναφέρον λοιπόν είπε ότι δεν θα παρευρεθεί, ε, δίνουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Πάολο Ντασίλβα και τον Αντρές ε, Κόμπε. Δεν ξέρω ποιος θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με την απάντηση και την ενημέρωση για την αναφορά 2553 του 2004 που μιλάει για την απαγόρευση των νανοσωματιδίων και την άλλη σχετικά με τα μικροπλαστικά βάσει της αρχής της ε, ε, πρόληψης για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η απάντηση της Επιτροπής δόθηκε το 2016. στις αρχές της προφύλαξης. Ε, όσον αφορά στα νανοσωματίδια, είναι νάνο υλικά που είναι σε μέγεθος ε, λιγότερο από 100 ε, νανό μέτρα και αυτά ήδη έχουν αντιμετωπιστεί το 2012 από το Ινκομισιόν βάσει μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης σχετικά με το κατά πόσο είναι κατάλληλο το ρυθμιστικό σύστημα. Έχουν βρεθεί τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εντός του συστήματος ε, και πρέπει να γίνει ένα tuning, ένα, μια καλύτερη προσαρμογή ας πούμε της νομοθεσίας στην αντιμετώπιση του θέματος των νοσοματιδίων και νοηλικών. η Κομισιόν έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές ε, στα κείμενα που ασχολούνται με τα χημικά, συγκεκριμένα την νομοθεσία για τα χημικά. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις ε, που διασφαλίζουν ότι η αξιολόγηση κινδύνου που γίνεται για οποιαδήποτε ουσία η οποία κατασκευάζεται, παρασκευάζεται, ε, εισάγεται σε νανομορφή ε, υπόκειται στη συγκεκριμένη νομοθεσία REACH ε, και ρυθμίζεται από αυτήν. Είναι ο κανονισμός του 2018. 181 που εγκρίθηκε το πέρυσι τον Δεκέμβρη και ξεκίνησε να ε, είναι σε ισχύ από τον ε, Γενάρη του, θα ξεκινήσει να είναι σε ισχύ από τον Γενάρη του 2020 Έχουμε κάποιες χημικές ουσίες που έχουν καταχωριστεί ήδη και πρέπει να ε, δούμε τον τοσχέ που τις αφορά, να δούμε αν υπάρχουν ε, νανοηλικά και αν υπάρχει συγκεκριμένη πληροφόρηση σχετικά με αυτά. Αυτές οι αλλαγές μαζί με τις συγκεκριμένες ε, απαιτήσεις βάση της νομοθεσίας για άλλα υλικά, όπως ας πούμε τα καλλιντικά, τα τρόφιμα κτλ όπως διαπιστώνει η Κομισιόν, μας δίνουν την απαραίτητη κάλυψη έναντι των δυνητικών κινδύνων που ε, προκύπτουν από την παραγωγή νανοηλικών. Φυσικά θα υπάρχει μια αναθεώρηση του κανονισμού REACH μετά το 2020 και της εφαρμογής του, όπως ε, θα προκύψει στην πράξη. Τώρα για τα μικροπλαστικά που είναι σωματίδια μικρότερα από τα 5 νανόμετρα και περιλαμβάνουν πολυμερή. Υπήρξαν αντικείμενο έντονη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Κομισιόν πολλά χρόνια είχε δράσει στον τομέα αυτό προσπαθώντας να συλλέξει πληροφορίες ε, για να μπορέσει να λάβει αποφάσεις με βάση μια ενημερωμένη ας πούμε και περιστατωμένη άποψη. Τα μέτρα διαχείρισης έχουν να κάνουν ε, με την ε, παραγωγή μικροπλαστικών που παράγονται και υπάρχουν στο περιβάλλον και επηρεάζουν το περιβάλλον και τους ανθρώπους ε, γιατί ε, προκύπτουν από τα προϊόντα που τα περιέχουν. Τα μικροπλαστικά υπάρχουν ε, στο περιβάλλον ούτως ή άλλως, χωρίς να υπάρχει πρόθεση, αλλά υπάρχουν και 6.000 τόνοι που οι θελημένα απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Αυτά θα αντιμετωπιστούν μέσα από τις ε, περιορισμούς που θα ετοιμάσει το Ευρωπαϊκό, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών ε, κατόπιν επιταγής της Κομισιόν. Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου θα είναι σε δημόσια διαβούλευση και μετά αυτός ο φάκελος με τους περιορισμούς θα συζητηθεί στις διάφορες επιτροπές όπως την ΕΟΚ και την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων με σκοπό οι γνωμοδοτήσεις ε, να έρθουν σε μας ε, μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους και εμείς στη συνέχεια με βάση αυτές να προτείνουμε περιορισμούς για την ηθελημένη απελευθέρωση μικροπλαστικών. Αυτή η θελημένη απελευθέρωση μικροπλαστικών ήδη με έναν γενικότερο τρόπο περιέχεται στην υφιστάμενη νομοθεσία που μιλάει για, τα, ε, για άλλες ε, ουσίες όπως ε, τα πετρελοειδή. Υπάρχουν διάφοροι τομείς φυσικά που μπορούν να συμπεριληφθούν, ειδικά αυτοί που αναφέρονται στις αναφορές, π.χ. τα λοιπάσματα. Μπορεί να έχουμε περιτυλίγματα, ας πούμε, που περιλαμβάνουν μικροπλαστικά και όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν στον κατάλληλο κανονισμό αλλά και με μονομένα ανατομέα ε, αυτή τη στιγμή καλύπτονται ας πούμε μόνο τα καλυπτικά, αλλά μπορούμε να έχουμε και τα λοιπάσματα και άλλα γεωργικά προϊόντα, όπως τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σπόρους. Όλα αυτά θα πρέπει να μπουν στην διαδικασία αυτή του περιορισμού και να σας πω ότι αυτή η διαδικασία είναι αυτή τη στιγμή να εξελίξει και δίνω το λόγο και στο συνάδελφο για να σας πει κάποια πράγματα σχετικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες για την έκφραση της ανησυχίας τους. Η στρατηγική για τα πλαστικά που παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2018 αντιμετώπισε ειδικά το πρόβλημα των μικροπλαστικών και τις ανησυχίες των πολιτών αλλά και των επιστημόνων. Όσον αφορά τα προβλήματα που προκαλούν τα μικροπλαστικά. Η Κομισιόν έχει δείξει την πρόθεσή της να αντιμετωπίσει το θέμα των μικροπλαστικών μέσα από τη στρατηγική για τα πλαστικά. Και αυτά που ε, απελευθερώνονται, στο περιβάλλον ηθελημένα και αυτά που απελευθερώνονται μη ηθελημένα, αυτά που δεν είναι ηθελημένα εκεί, όπως ας πούμε στην υφαντουργία, ή ε, ε, συσκευασία συσκευασίες για την προστασία των ε, διαφόρων φαρμάκων. Αυτά είναι πράγματα που δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή. Αναφέρονται στις αναφορές και η Κομισιόν έχει αναλάβει δράση σε αυτό τον τομέα, ξεκινώντας με τη συμφωνία σε επίπεδο διαφόρων τομέων της βιομηχανίας, ε, π.χ. της εφαντουργίας. Ήταν μια θελούσια συμφωνία επί των μεθόδων παρακολούθησης της παραγωγής και συμπερίληψης μικροπλαστικών στα προϊόντα εφαντουργίας. Υπήρξε και συνεργασία με την υπηρεσία προτυπών και τυποποίησης για να βγουν συγκεκριμένα πρότυπα για τα μικροπλαστικά. Επίσης, η αναθεώρηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό που ολοκληρώθηκε η πρώτη της ανάγνωση πρόσφατα ήδη προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη υπό συγκεκριμένε συνθήκες θα παρακολουθούν την ύπαρξη μικροπλαστικών στο πόσιμο νερό. Επίσης υπάρχει και το refit της ε, οδηγίας ε, των ε, περί απορριμμάτων και λιμάτων. Και εκεί αναφέρονται τα προϊόντα υφανουργίας. Αυτό είναι ακόμα ένα εξέλιξη. Θα λάβουμε υπόψη μας λοιπόν και το Κοινοβούλιο και τα όσα αναφέρουν οι αναφέροντες Επίσης υποστηρίζουμε την έρευνα. Υπάρχουν πολλά project που χρηματοδοτούνται μέσα από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίντερεκ για τα μικροπλαστικά, το Mark Mermaids. Επίσης όλα αυτά είναι προσπάθειες να βρεθούν λύσεις για το πώς να αποφύγουμε την απελευθέρωση μικροπλαστικών. Επίσης, ε, οι μονάδες επεξεργασίας λιμάτων ε, είναι υποχρεωμένες να έχουν φίλτρα που θα συλλέγουν τα μικροπλαστικά και δεν θα ρηπαίνονται τα ύδατα. Όλα αυτά είναι τεχνολογίες που αυτή τη στιγμή εξετάζονται. Αλλά όπως και να έχει, η Κομισιόν προτιμά λύσεις που είναι πιο ψηλά στην ε, ε, αδελισίδα αξίας. Δηλαδή πράγματα που έχουν να κάνουν με το τέλος της διαδικασίας, ε, αν υπάρχει συγκεκριμένο κόστος, θα πρέπει να δούμε ποιος θα συμβάλλει, το κράτος ή οι εταιρείες που παράγουν τα μικροπλαστικά. Θα ξεκινήσει λοιπόν μια μελέτη του χρόνου ακριβώς ε, για τις τεχνικές λύσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν ε, να αποφύγουμε τα μικροπλαστικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τα μέλη της Επιτροπής τώρα. Ποιος θέλει το λόγο. Ο κύριος Σαλίβα. Καταρχά να ευχαριστήσω του αναφέροντες για αυτή την ε, πάρα πολύ σημαντική παρουσίαση του θέματος. Είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και το εκφράζουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες. Το καλύτερο για το θέμα αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σύγκληση από όλα τα πολιτικά κόμματα ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προσπάθεια που πρέπει να γίνει προκειμένου να ε, προστατεύσουμε το κλίμα. Το θέμα των πλαστικών είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι η παραγωγή και η χρήση του είναι το επίκεντρο, στο επίκεντρο κριτικών πολλών πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο να γίνει μια κρόαση επί του θέματος ε, στις αρχές του 2020. Από πλευρά ε, θεσμικών οργάνων έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά. Ε, υπάρχει και δουλειά σε εξέλιξη. Το Σεπτέμβριο οι Ευρωβουλευτέ ενέκριναν τη στρατηγική του ε, και θεωρούν ότι πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση των πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι το 2030 όλες οι πλαστικές συσκευασίες θα είναι ανακυκλώσιμες. Επιπλέον, Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει απαγόρευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ε, εξαλείψουμε τη συσσόρευση πλαστικών, ε, κυρίως σε προϊόντα όπως καλλιτικά και απορριπαντικά μέχρι το 2030. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να ληφθούν μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η χρήση μικροπλαστικών ε, σε κλωστοϊφαντουργία, σε μπογιές κλπ. Επίσης ζητήθηκε να μειωθεί η ε, χρήση πλαστικών ε, που φτάνουν ε, στην ε, ε, θάλασσα και δεν υπάρχει αντίστοιχη χρήση άλλου υλικού σε σχέση με τα πλαστικά. Επίσης, συμβατικά πλαστικά, τα οποία εύκολα σπάνε σε πολύ μικρά κομματάκια λόγω των πρόσθετων ουσιών και συμβάλλουν στην ρήπανση μικροπλαστικών των ωκεανών. Γι' αυτό ακριβώ είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αναφορές αυτές να παραμείνουν ανοιχτές. Ο κύριος Γιάρ. Äh, Έχετε πολύ σωστά διατυπώσει την κατάσταση. Είπατε ότι πρέπει μαζί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Ε, πρέπει και αυτοί να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Καλό είναι η Επιτροπή μας πάντοτε να συνεργάζεται με την υπεύθυνη ειδική Επιτροπή για να μπορέσουμε να έχουμε και μια πολιτική επίπτωση μεγαλύτερη. Να ενημερώσουμε και τον αναφέροντα ώστε να γνωρίζει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο Υπάρχει πολλή δουλειά που γίνεται σε επίπεδο νανοσωματιδίων και μικροπλαστικών. Κρατάμε λοιπόν ανοιχτή την αναφορά και προχωράμε στο επόμενο στάδιο Επιτροπή σε αυτό το θέμα. Τέλεια. Επειδή δεν υπάρχει κάποιο άλλο, ο οποίο θα ήθελε το λόγο, η πρόταση της Προεδρίας είναι να παραμείνει ανοιχτή να παραμείνουν μάλλον ανοιχτέ αυτέ οι αναφορές ε, κατόπιν των όσων είπαν και ευρωβουλευτέ, να ζητήσουμε επικαιροποιημένε πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών υδάτων και τη συνέχεια τη διάσκεψη των ενδιαφερομένων μερών ε, που έγινε τον Νοέμβριο του 2018. Να παρακολουθήσουμε επίση και την εφαρμογή τη στρατηγική για τα πλαστικά και την οδηγία για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου συγκεκριμένων προϊόντων πλαστικού και μετά από ε, όσα ακούσαμε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Βάντερ Λάιον, ότι ε, θέλουμε να απαγορεύσουν τα πλαστικά μιας χρήσης, θα παραμείνει ανοιχτή αναφορά ε, λόγω της σημασίας τους. Ε, επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι η Προεδρία συμφωνεί να γίνει κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημοσίας Υγείας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε την ουσία του θέματος. Αυτή είναι η πρόταση της Προεδρίας. Ωραία. Τέλεια, ολοκληρώνεται το σημείο αυτό. Και τώρα είμαστε στο σημείο 14, αλλά μισή ώρα νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν ε, να ξεκινήσει η συγκεκριμένη αναφορά. Δεν υπάρχει παρουσία των αναφερομένων και μας είπαν ότι δεν θα έρθουν. Βλέπω ότι ο κύριος Ντασίλβα ούτως ή άλλως είναι εδώ και θα απαντήσει αυτός πάλι στη συγκεκριμένη αναφορά. Αν ε, συμφωνούν οι συντονιστές των ομάδων, μπορούμε να συνεχίσουμε με την ε, αναφορά αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ε, πολιτική ομάδα που ξέρει ότι υπάρχει κάποιος βουλευτής ο οποίος ε, θέλει να είναι παρόν για να παρουσιάσει τα επιχειρήματά του για το θέμα αυτό και ίσως εμείς προχωράμε και μπορεί να βρεθεί κάποιος ευρωβουλευτής ο οποίος δεν μπορέσει να λάβει το λόγο και μετά πει στην Προεδρία κοιτάξτε και ξεκινήσετε μισή ώρα νωρίτερα την αναφορά και εγώ δεν ήρθα εγκαίρως. Το λέω γιατί όπως έχουμε διαμορφώσει την ημερήσια διάταξη και οι ε, βουλευτές ξέρουν ακριβώς πότε ξεκινάει η αναφορά τους, ε, ε, θα στερήσουμε δικαιώματα σε κάποιο βουλευτή. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συντονιστές που είναι παρόντες στην αίθουσα τι άποψη έχουν. Να κάνουμε διάλειμμα και να ξεκινήσουμε στις παραπέντε για να μην χαθεί κάποιος βουλευτής ο οποίος θα ήθελε να παρέμβει ή να συνεχίσουμε, μιας και ο αναφορών δεν θα έρθει και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής είναι παρόν. Uh, Ο Conrado Matza είναι εδώ. Άρα είναι και εδώ ε, και οι δύο. Συνεχίζουμε. Ωραία. Okay. Ωραία. Θα κάνουμε διάλειμμα, αν δεν κάνω λάθος, στο επόμενο, διότι εκεί έχουμε παρουσία του αναφέροντος. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την αναφορά. Αναφορά 349 του 2018 από Γερμανό υπήκο εξ ονόματος Intentions Media Minds για την εφαρμογή νομοθεσία σχετικά με τη χρήση πλαστικών. Αναφορά επίσης 191 του 2018 Γερμανού υπηκόου σχετικά με τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων και αναφορά 758 του 2018 από Βρετανό υπήκο σχετικά με την παραγωγή πλαστικών και τη βελτίωση της κυκλικής οικονομίας. Επειδή λοιπόν οι αναφέροντες είπαν ότι δεν θα παραβρεθούν, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντασίλβα εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους αναφέροντες για τις ανησυχίες που εξέφρασαν ζητούν τη δράση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, η 0191 ε, θεωρεί ότι δεν έχουν πάρθει αρκετά νομικά μέτρα ε, εμείς όμως πιστεύουμε ότι η Επιτροπή βρίσκεται στο σωστό δρόμο γιατί η στρατηγική για τα, για τα πλαστικά έχει θέσει ε, στόχο ε, για τον ε, βιώσιμο στόχο για τον τομέα των πλαστικών να είναι πιο ανταγωνιστικός και πιο βιώσιμος και αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο το ζήτημα της θαλάσσης ρήπανσης από τα πλαστικά. Οι εφαρμοστικές δράσεις που έχουν ληφθεί αναφορικά με την στρατηγική των πλαστικών έχουν να κάνουν ακριβώς με την ρήπανση των πλαστικών. Θυμάστε την ε, παγόρευση στα μικροπλαστικά, όπως αναφέρθηκε, αλλά και την ε, οδηγία για, την, ε, για τον εξοπλισμό ψαρέματος και την χρήση πλαστικών μιας χρήσης. Αυτή η οδηγία θέτει φιλόδοξους στόχους σε διαφορετικούς τομείς. Ε, ε, θα αναφέρω, επί παραδείγματι, το στόχο για ε, να μαζευτούν τα πλαστικά μπουκάλια μέχρι το 2029 και την ανακύκλωση κατά 25% μέχρι το 2025 των πλαστικών μπουκαλιών Κάποια προϊόντα έχουν απαγορευθεί γιατί υπάρχουν ε, βιώσιμα εναλλακτικά μέσα για να τα αντικαταστήσουν. Ε, επομένως, ε, θεωρούμε ότι η εφαρμογή της οδηγίας πηγαίνει στο σωστό δρόμο. Εμείς Αναφερόμαστε επίσης και, στο, και στην ανακύκλωση του, προϊόν, του, του περιεχομένου. Έχουμε και εκεί ε, φιλόδοξους στόχους. Ο στόχος είναι 10 εκατομμύρια ανακυκλωμένου, ανακυκλωμένου πλαστικού σε νέα προϊόντα μέχρι το 2025. Συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Ε, όπως ξέρετε, 20 του μηνός ε, θα παρουσιαστούν ε, οι συμβιβασμοί από τη συμμαχία του, του πλαστικού για το πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να ε, υλοποιήσουμε αυτό το στόχο είναι σημαντικό όχι μόνο για τη βιομηχανία, όχι μόνο για την ε, μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ε, γιατί η ανακύκλωση είναι καλύτερη, καλύτερη μέθοδος από την παραγωγή, σχετικά με, συγκριτικά με την παραγωγή ε, σχετικά με την παραγωγή από ε, πρώτες ύλες, αλλά γιατί εν γέννη προστατεύει το περιβάλλον. Αυτά τα φιλόδοξα μέτρα λοιπόν ε, θα είναι σημαντικά και έναν άλλο λόγο γιατί χώρες ανά τον κόσμο ακολουθούν το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες χώρες ήδη έχουν ε, προετοιμάσει ή υιοθετήσει στρατηγικές κατά το πλαστικό. Άλλες χώρες ε, έχουν πάρει μέτρα για την χρήση των πλαστικών μιας χρήσης. Ο Καναδάς, για παράδειγμα, παρουσίασε την πρόταση, του, ε, την πρόταση νόμου για την ε, χρήση πλαστικών μιας χρήσης, κατά το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, εμείς θέτουμε, ε, το, θέτουμε τα πρότυπα που ακολουθούνται από χώρες ε, ανά τον κόσμο, So the Basel Convention has taken action on plastic. Η UNEP έχει επίση παρουσιάσει μια διακήρυξη για την χρήση πλαστικών μια χρήση. Ευχαριστούμε πολύ. θα αναφερθώ στο σημείο 15 της ημερήσιας διάτασης ε, και την αναφορά 0758 Επομένως, ε, θα παρέμβω μετά για αυτά τα ζητήματα. Okay, let's do it in the next. Ωραία, τότε να γίνει στην επόμενη αναφορά. Τέλεια. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος. I am sorry, I'm sorry. Α, συγγνώμη. Υπάρχει κάποιος από την Επιτροπή ο οποίος ε, θέλει να πει κάτι για τη συγκεκριμένη αναφορά. Ο κύριος Γιάρ. Το μόνο θέμα είναι αν θα το αφήσουμε ανοιχτό ή θα το κλείσουμε. Από τη μία είναι ότι υπάρχουν τόσες πολλές πρωτοβουλίες ε, που έχει πάρει η Κομισιόν. Παγκασμίως ε, υπάρχουν συμφωνίες. Μπορεί ό,τι κάνει θέλει κανείς να κάνει, είτε να την κλείσει είτε να την ανοίξει από τον πρόεδρο εξαρτάται. Είστε η αρχηγός αυτής της διαδικασίας. Συμφωνώ με τον συνάδελφο, πολλά έγιναν, πολλά έχουν μπει σε σειρά για να γίνουν, αλλά ποτέ τίποτα δεν είναι αρκετό όταν μιλάμε για το κλίμα και τη μείωση των πλαστικών. Οπότε... Λοιπόν, η πρόταση της Προεδρίας λαμβάνοντας υπόψη ε, και το σύνολο των μέτρων που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια για τη βιώσιμη χρήση πλαστικών και την παραγωγή πλαστικών, για την αντιμετώπιση των ε, βιώσιμης χρήσης των πόρων και των ε, πλαστικών αποβλήτων και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηγέτης σε αυτή τη μεγάλη μάχη που γίνεται και βλέποντας και την προηγούμενη της αναφοράς, η πρόταση της Προεδρίας είναι να ολοκληρωθεί η εξέταση της συγκεκριμένη αναφοράς, εάν συμφωνείτε κι εσείς. Ωραία. Ωραία, να περάσουμε στην επόμενη αναφορά. Μου είπαν ότι είναι εδώ ο αναφέρον. Η επόμενη αναφορά είναι η 1013 του 2018 του Αλεσάνδρο Τζοβανέτη, η Ιταλική Ιθαγένεια, σχετικά με τη χρήση ενό μόνο υλικού στη συγκευασία προϊόντων σούπερ μάρκετ. Και επίση την αναφορά 82 του 2019 τη Έλενα Μιχαέλα Μπλέτια, Ρουμανική Ιθαγένεια, σχετικά με την καλύτερη χρήση των πλαστικών συσκευασιών. Ο αναφέρον, ο κύριος Αλεξάνδρο Τζοβανέτη, είναι παρόν. Νομίζω ότι έχετε φέρει και μια παρουσίαση PowerPoint. Η παρουσίαση πρέπει να γίνει σε πέντε λεπτά. Έχετε πέντε λεπτά για να κάνετε την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, αξιότιμη επιτροπή, σας ευχαριστώ που δέχεστε την αναφορά μου. Όπως γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρωτοπόρος στην ε, παγκοσμίω για την εφαρμογή νομοθεσίας για το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Η τελευταία απόφαση για τα πλαστικά είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αλλά τι θα γίνει σε ένα ευρωπαϊκό κράτο για τη μείωση των αποβλήτων και την ε, αύξηση τη ανακύκλωση. Κάθε κράτο μπορεί να αποφασίσει για τον κύκλο ζωή των αποβλήτων και επίση οι επιχειρήσει εφαρμόζουν ε, την νομοθεσία με το δικό του τρόπο και μόνον. Η συσκευασία ε, είναι ακόμα πολύ σοβαρό θέμα στι μεγάλε αλυσίδε σούπερ μάρκετ και τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Γι' αυτό ζητώ από όλου εσά να παρέμβετε για να αλλάξουν τι συσκευασίε ξεκινώντα από τι μεγάλε επιχειρήσει. Θα μπορούσε να αλλάξει η συσκευασία ε, χρησιμοποιώντας ε, ως γνώμονα το σχήμα ή τη χρήση ενός προϊόντος. Επίσης ε, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ και έτσι και οι καταναλωτές να επιλέξουν. Σε περίπτωση αναλώσιμων τροφίμων μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικές συσκευασίες για να προστατεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης όλες οι οδηγίες θα πρέπει να είναι ενιαίες σε όλη την Ευρώπη και να χρησιμοποιούνται εύκολα σήματα για άτομα όλων των ηλικιών, ώστε να αυξηθεί η ανακύκλωση και να ε, μην γίνονται λάθη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε στην πρώτη διαφάνεια. Για παράδειγμα, παιδικά κέικ. Ε, από τη μεγάλη κλίμακα διαμονή έχουμε το χαρτοκιβώτιο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα κέικ. Τα κέικα είναι σε πλαστικέ συσκευασίε. Και μετά υπάρχουν χαρτοκιβώτια και πάλι. Και μετά ε, ο περιτύλιγμα για τα κέικ. Επομένω, ε, για κάτι το οποίο θα καταναλώσουμε σε δύο λεπτά, έχουμε πάρα πολύ πλαστικό και χαρτί τα οποία πηγαίνουν χαμένα. Ε, ο καθένα μπορεί να καταλάβει ποια από αυτά τα υλικά είναι απαραίτητα και ποια είναι ασφαλή και ανακυκλώσιμα σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να βρούμε την κατάλληλη λύση. Ε, αυτά τα σήματα πολύ συχνά εμφανίζονται σε συσκευασίε, σε κονσέρβες και διάφορα προϊόντα. Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά όλα τα υλικά κάποιο πριν τα πετάξει και αυτά είναι κακά παραδείγματα για σχεδιασμό συσκευασιών και ορισμένες φορές επηρεάζουν και το συνολικό κόστο ενός προϊόντος ε, που συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη. Αν η μητέρα φύση γνώριζε ότι βάζουμε φρέσκα φρούτα μέσα σε πλαστικές συσκευασίες, ε, δεν ξέρω τι θα έκανε, είναι απίστευτο. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε δύο διαφορετικές πλαστικές φιάλες νερού. Έχουμε τον ίδιο χρώμα, αλλά δύο διαφορετικές ε, ε, δυνατότητες πάχους πλαστικού και δύο διαφορετικές τιμές. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν πληρώνουμε για το προϊόν ή για τη συσκευασία. Ε, ζητώ να δεχτείτε την αναφορά μου για να επιταγχυθεί η διαδικασία σε όλες τις χώρες μέλη και να μειώσουμε τα πλαστικά. Ε, σας παρακαλώ να τα διευκολύνουμε όλα αυτά γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς στον κύριο Λεωνάρδο Μάτσα και έχουμε και τα σχόλια για την 758 του 2018. Μας είπατε ότι θα μιλήσετε και για αυτήν, ε, την οποία την ε, αναβάλατε προηγουμένως για να μιλήσετε για το θέμα αυτό, μαζί με τις άλλες δύο αναφορές. Yes, indeed, my... Η παρέμβασή μου όντω αναφερόταν σε αυτές τις τρεις αναφορές, ε, συμπεριλαμβανομένης ε, της ε, τελευταίας από, προηγούμενο, το προηγούμενο σημείο. Ευχαριστώ για το, το Προεδρείο που μου δίνει το λόγο. Αναφορικά λοιπόν με αυτές τις τρεις αναφορές που σχετίζονται με την πρόληψη ε, πρόληψη ε, ρήπανσης που δεν χρειάζεται και την καλύτερη διαχείριση ε, των πλαστικών συσκευασιών, οι στόχοι έχουν ε, σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ε, αλλά και με ε, εξελισσόμενες πρωτοβουλίες. Μία πρωτοβουλία κλειδί που αναφέρθηκε μάλιστα και σε σχέση με προηγούμενες αναφορές είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Πλαστική Κυκλική Οικονομία που υιοθετήθηκε το 2018 τον Ιανουάριο Μέχρι το 2030 όλα τα πλαστι... όλη η πλαστική συσκευασία θα πρέπει να ε, είτε να ανακυκλώνεται είτε να ε, επαναχρησιμοποιείται με έναν οικονομικό τρόπο. Αυτός ο στόχος θα υλοποιηθεί ε, μέσα στο ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο ένα κέριο εργαλείο που υπάρχει από το 1994 είναι η οδηγία για, το, για τη συσκευασία που είναι το πρώτο μέτρο για την ε, ε, πρόληψη κατά της περιτής, ε, των περιττών συσκευασιών. Πέρσι αυξήθηκαν οι στόχοι ανακύκλωσης για διάφορα υλικά, συμπεριλαμβανομένου και του πλαστικού. Ο στόχος εκεί διπλασιάστηκε και αναφορικά σε σχέση με τα σημεία αυτά, στην τελευταία αναθεώρηση η Επιτροπή εξέτασε το κατά πόσο θα είναι ε, εφικτό να ε, ενισχυθούν ε, οι απαιτήσει για τις πλαστικές συσκευασίε που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν προκειμένου, σκεπτόμαστε την, την υψηλής ποιότητας ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους. Αυτές λοιπόν είναι βασικές απαιτήσει που έχουν θεσμοθετηθεί μέχρι στιγμής για την ενίσχυση του, της ανακύκλωσης των συσκευασιών. Εξετάζουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή πώς αυτές οι απαιτήσει της οδηγίας μπορούν να ε, ενισχυθούν και η Επιτροπή θα ε, αποφασίσει για την αναθεώρηση αυτών των απαιτήσεων και ίσως ε, θέση και πρόταση μέχρι το τέλος του 2020. Ένας εκ των αναφερόντων ε, εξέφρασε την ε, ανάγκη για την καλύτερη ετικετικοποίηση για το, που θα βοηθήσει τους καταναλωτές πώς να πετάν τα, τα προϊόντα της συσκευασία. Η οδηγία της συσκευασία Κατευθύνει λοιπόν ε, τους, ε, το πώς θα αναγράφονται πληροφορίες ώστε, να, ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ε, επιστρέψουν τις συσκευασίε, αλλά και τον ρόλο που έχουν οι καταναλωτές στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των συσκευασιών. Ένα άλλο εργαλείο που πρέπει να αναφερθεί σχετικά με τη βελτίωση της, του σχεδιασμού των συσκευασιών Πιστεύουμε ότι θα, θα δώσει μάλιστα και καρπούς. Ήταν η προηγούμενη αναθεώρηση όπου ε, ρύθμιζε την, ε, το ποσό που θα πλήρωναν ε, οι παραγωγοί για την λήξη του προϊόντος για παράδειγμα, θα πρέπει να δουν κατά πόσο είναι εύκολο να ανακυκλωθεί. Σε αυτή λοιπόν την ε, τροποποίηση η Επιτροπή ετοιμάζει οδηγίες στα κράτη-μέλη, θα είναι διαθέσιμη στο τέλος του χρόνου. Μια άλλη πρωτοβουλία που υπερβαίνει τον τομέα των συσκευασιών, αλλά επίσης ε, σχετίζεται στο πλαίσιο της ανακυκλωσιμότητας, είναι ε, η η Συμμαχία για, την, για τα κυκλικά πλαστικά που οργάνωσε η Επιτροπή με, με ε, το, φορείς από τον ε, κύκλο ζωής των πλαστικών υιοθέτησε μάλιστα και μία διακήρυξη όπου παρουσίασαν ε, το στόχο τους για το μέλλον και τη δέσμευσή τους για δράση. Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτή την, ε, ε αυτή την ε, κατάσταση παρέχοντας ε, ε κατευθυντήρες γραμμές για την ανακύκλωση των πλαστικών. Κατακλείδη, οι προτάσεις των αναφερόντων έχουν ληφθεί υπόψη τους και τις, και τις έχουμε εξετάσει. Το πλαίσιο πολιτικής έχει γίνει ε, καλύτερο στο να δίνει κίνητρα ε, στη, στον τομέα των συσκευασιών. Έχουν, δώσει, έχουν δοθεί μάλιστα κατευθυντήρες γραμμές ε, για, το κόστος της συσκευασίας και σε αυτό το τομέα εργασίας πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν περισσότερες, περισσότερα κίνητρα στο μέλλον για την βελτίωση της πρόληψης της, ε, των αποβλήτων. As Όπως ανέφερε η Επιτροπή, λέει ο κ. Σαλίβα, ε, ε, όλα τα προβλήματα Όλα τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται όμως το πρόβλημα εν μέρη ε, αντιμετωπίζεται και υπάρχει σύγχυση μεταξύ των πολιτών. Υπάρχει ο τομέας ε, της ανακύκλωσης, διάφορα πλαστικά μπαίνουν στην αγορά. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή ενώπιν της Επιτροπής η συγκεκριμένη αναφορά. Ευχαριστώ. Κυρία Εύη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια αναφορά η οποία θα πρέπει να μείνει ανοιχτή και γιατί ε, εφιστά την προσοχή σε ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη φιλοδοξία και μονίμω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάλυση τη μα είπε για τι διάφορε πρωτοβουλίε ε, οι οποίε ε, θα ξεκινήσουν του επόμενου μήνε, ε, όπω για παράδειγμα την αναθεώρηση των απαραίτητων στοιχείων για τι συσκευασίε και την ευθύνη των παραγωγών. Επομένω, τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την οδηγία. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε καθήκον να προσέξουμε ιδιαίτερο στο θέμα αυτό, διότι το να μειώσουμε σήμερα τη χρήση των πλαστικών σε μια μακρά σειρά από είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη έχει κάνει ε, σημαντικά βήματα και θεωρούμαστε και πρωτοπόροι στον τομέα και μας ακολουθούν άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά είναι εξίσου αληθές ότι ε, τα ίδια θετικά βήματα δεν είναι ε, η λύση του προβλήματος. Όπως για παράδειγμα οι πλαστικές φιάλες για το νερό, όπου δεν υπάρχουν ε, μεγάλη μεγάλοι θαραλέοι στόχοι μείωσης της χρήσης πλαστικών. Πιστεύω ότι πρέπει λοιπόν και μπορεί να παραμείνει ανοιχτή αφορά αυτή για να αναθεωρήσουμε στο μέλλον και το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Έχει κάποιον άλλον ο οποίος θέλει να ζητήσει το λόγο από το ΕΛΚ για παράδειγμα. Όχι. Θα ήθελα να δώσω δύο λεπτά λοιπόν το λόγο στον αναφέροντα για να σχολιάσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αν θέλετε. Ναι, ναι, φυσικά. Ναι, όντως, ευχαριστώ πολύ. Βλέπω, όπως είπατε, ότι ακόμα δεν έχουμε εστιάσει σε αυτό. Έχετε πολλή δουλειά ακόμα να κάνετε για να, κάνετε, για να προχωρήσετε το θέμα των αποβλήτων. Ήρθα σήμερα εδώ και δεν περίμενα ότι στο Βέλγιο δεν κάνουν καθόλου ανακύκλωση. Αν πας σε ένα μπαρ θα δεις ότι τίποτα δεν ανακυκλώνουν. Περίεργο λοιπόν. Δεν ξέρω γιατί κάθε χώρα δεν ακολουθεί τη βασική κατεύθυνση που δίνει η Ευρώπη.

Η πρόταση της Προεδρίας, μετά από όσα ακούσαμε από τον αναφέροντα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη ενέκρινε σχετικό ψήφισμα στις 13 Σεπτεμβρίου του 2018 για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά και μια κυκλική οικονομία, αλλά μετά από όσα ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μας λέει ότι πρέπει να συνεχίσει η αναθεώρηση των απαιτήσεων του σχεδιασμού των συσκευασιών και λαμβάνοντας υπόψη και το πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ε, θα παραμείνει ανοιχτή και ε, θα παρακολουθήσουμε την εφαρμογή της στρατηγικής για τα πλαστικά και τις οδηγίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου ε, συγκεκριμένων πλαστικών προϊόντων στα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η πρόταση της Προέδρου. Αν συμφωνείτε όλοι, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Πρόκειται για την αναφορά 1124-2018 από Πολωνό Υπήκο που φέρει άλλες δύο υπογραφές σχετικά με την καλή διαβέωση των μελισσών. Ο αναφέρον δεν μπορεί να παρευρεθεί ε, στη συνεδρίαση της Επιτροπής και γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κύριο ε, Ντενίς Σιμονίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω στα γαλλικά. Η επάντηση της Επιτροπής ε, έχει αρκετά σημεία που ε, καλύπτουν τις αρμοδιότητες. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μια περίληψη όλων αυτών λοιπόν. Για την ευζοία των μελισσών υπάρχουν συγκεκριμένα κείμενα. Η νομοθεσία για την ευζοία των, ε, ε, ε, των, των ζώων στιάζει κυρίως σε αυτά που έχουν σπονδυλική στήλη και έχουν κάποια, κάποιες μορφές συνείδησης. Υπάρχει μια συζήτηση επιστημονική για τα, για τα έντομα και αυτό φυσικά επαφίεται στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Δεδομένου αυτού λοιπόν υπάρχουν αρκετά μέτρα, ειδικά μέτρα, ε, που υπάρχουν ε, σε διαφορετικές πολιτικές, ε, όπως για παράδειγμα η κοινή αγροτική πολιτική, όπου υπάρχει η δυνατότητα εθνικών πλάνων για τους, για τους μελισσοπαραγωγούς, που σχετίζονται με τη συγχρηματοδότηση της προστασίας των μελισσών και περιλαμβάνουν την ε, διαχείριση αλλά και, το, και, την, τη διατήρηση και τη συντήρηση των μελισσών. Όπως σας είπα, αυτά είναι συγχρηματοδοτούμενα με την Ένωση. Επίσης, στα πλαίσια της ε, ΚΑΠ υπάρχει ένας πιο οριζόντιος ε, τρόπος για την προστασία των μελισσών, κυρίως στον τομέα του, του πρώτου πυλώνα, ε, για την προστασία των ε, μόνιμων γεωργικών εγκαταστάσεων και της ε, βιοπικιλότητας, για στην προστασία της βιοπικιλότητας. Υπάρχουν λοιπόν κάποια μέτρα που ευνοούν το βιότοπο των μέλισσών, όχι μόνο για τις οικόσιτες μέλισσες, αλλά γενικά για τις μέλισσες. Υπάρχουν επίσης δευτερευόντως μέτρα στα πλαίσια της αγροτικής ανάπτυξης που επίσης μπορούν να ε, δώσουν ε, ε, βοήθεια στους, στον τομέα των μελισσών. Υπάρχουν επίσης περιβαλλοντικές πολιτικές. Ένα, μια, μια πρωτοβουλία που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2018 για τους επικολαστές ε, εστίαζε κυρίως ε, τις, ε, τις μέλη μέλητες αλλά όχι μόνο για, τον για την εκλογήκευση της χρήσης των των εντομοκτώνων. Το πρόβλημα των επικονιαστών είχε αντιμετωπιστεί με αυτό το για, εν κατακλείδη, η Γενική Διεύθυνση Υγείας ε, έχει δώσει μέτρα για τις ασθένειες των μελισσών, για, σχετικά μάλιστα με την εισαγωγή ε, ασθενειών από, άλλα, από, από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ανταλλαγής μελισσών μεταξύ κρατών μελών. Εντάχει, λοιπόν, αυτά είναι τα μέλη που έχουν ληφθεί από τις ε, ε, που έχουν ληφθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μέλισσες και των ε, επικονιαστών. Όσον αφορά τώρα στην ε, αναθεώρηση του ΚΑΠ, υπάρχουν ορισμένα μέτρα που για την ενίσχυση του τομέα των μελισσοπαραγωγών ή για την, για την προστασία των κατοίκων εν προκειμένου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Και τώρα ο λόγο στα μέλη τη Επιτροπής. Υπάρχει κάποιο ο οποίος θα ήθελε να λάβει το λόγο στο σημείο αυτό. Αν όχι, μετά από τα όσα ακούσαμε και διαβάζοντας και την αναφορά του αναφερομένου και ακούγοντας τα όσα μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μας λέει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ε, υπάρχουν κάποια ε, πιο γενικά μέτρα, αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο για τις μέλισσες και στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα μπορούσαμε ίσως να προβλέψουμε και μέτρα για την προστασία του κλάδου της μελισσοκομείας. Ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να παραμένει ανοιχτή η αναφορά, να αποσταλεί η αναφορά προς ενημέρωση στον Επίτροπο Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπέθρου, τον κύριο Χόγκαν ή στον επόμενο ε, αρμόδιο επίτροπο όταν θα συσταθεί η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσουμε και γνωμοδότηση από την Επιτροπή Άγκρη. Δεν ξέρω αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Αυτή είναι η πρόταση της Επιτροπής και μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη αναφορά. Η επόμενη αναφορά είναι η 611 του 2018 του Ισμαέλ Σάντσεφ Καστίγιο, Ισπανικής Ιθαγένειας, εξ ονόματος της Κομιτέ Προβιθιάν του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σεβίλης για την επιβολή δασμού των ΗΠΑ στην εισαγωγή όριμων ελιών από την Ισπανία. Ο αναφέρον είναι παρόν. Καλωσορίσατε λοιπόν και έχετε πέντε λεπτά για να μας παρουσιάσετε την αναφορά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά ο τομέας ε, των επιτραπέζιων ελιών, στην περιοχή της Σεβίλης ε, δίνει σε περίπου 10.500 άτομα θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ένα κλάδο ο οποίος είναι από τους κλάδους που πλήττονται, διότι οι εργαζόμενοι άνδρες και γυναίκες εδώ και χρόνια ε, υπόκεινται προστατευτισμό από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είναι εποχική εργασία και αυτή τη στιγμή πλήγονται και από τους δασμούς, τους δυσανάλογους που επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ ε, στις ε, επιτραπέζες ελιές, τις μαύρες ελιές. Το Υπουργείο Γεωργίας, όπως ξέρετε, έχει ζητήσει δασμούς οι οποίοι φτάνουν μέχρι και το 43,26% όσον αφορά τις μαύρες ελιές. Και αυτό σημαίνει ότι οι εξαγωγές της Ισπασίας ε, μειώθηκαν κατά 42,6% μεταξύ του Ιανουαρίου και του Νοεμβρίου του 2018 όσον αφορά του τόνους από 27,7 ε, ε, τόνους, ε, φτάσαμε στους 14,9 και τον Αύγουστο του 2018 οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 60% φτάνοντας από το 11,2 εκατομμύρια κιλά στα 240.000, δηλαδή 6,8 εκατομμύρια κιλά λιγότερα ουσιαστικά θα χαθεί ε, κατά πάσα πιθανότητα σταδιακά η όλη αυτή η αγορά οι εισαγωγέ από άλλες χώρες, από το Μαρόκο, από την Αίγυπτο, στο μεταξύ που έχουν αντίστοιχες όριμε ελιέ ε, ε, όπως και η Ισπανία, αυξήθηκαν κατά 25,7% από τα 3,4 πέρασαν στα 5,9 εκατομμύρια κιλά. Πρόκειται για δασμολογικά μέτρα τα οποία είναι άδικα και καταχρηστικά από πλευρά ΗΠΑ και δεν ε, καταφέρονται μόνο κατά τη επιτραπέζια ελιά τη Εβίλη, αλλά και κατά του συνόλου κοινή αγροτική πολιτική. γι' αυτό ακριβώ η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ζήτησε ο ΠΟΕ να συστήσει ένα πάλεν ε, για να εξετάσει την νομιμότητα αυτών των μέτρων ε, για την εισαγωγή των επιτραπέζιων μαύρων ελαίων της Ισπανίας. Έχει περίπου 1,5 χρόνο από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση στο πάνελ, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μακρά διαδικασία και το μεταξύ οι εργαζόμενοι άνδρες και γυναίκες της επαρχίας της Εβίλης και στην ε, αυτόνομη περιοχή της Ανδαλουσίας ε, πληρώνουν το τίμημα. Ε, μετά από αυτό το βήμα, οι Ηνωμένε Πολιτείε εξακολουθούν να λένε ότι οι επιδοτήσει τη κοινή αγροτική πολιτική, οι οποίε λαμβάνονται από του παραγωγού όριμων ελαίων, παραβιάζουν του κανόνε του ΠΟΕ. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πάρα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο για οποιαδήποτε άλλη χώρα η οποία θα έρθει να ανταγωνιστεί τα προϊόντα της Ένωσης ε, και λαμβάνονται επιδοτήσεις από την ΚΑΠ. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να οικειοποιηθεί το θέμα της υπεράσπισης ε, των ε, ελιών για τους δασμούς που επιβάλλονται από τη ΣΥΠΑ. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση πρώτου επίπεδου γιατί η κυβέρνηση Τραμπ δημιουργεί πραγματική ζημία στον κλάδο και στην ίδια την ΚΑΠ γιατί θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως υπάρχει ήδη σε όλο τον τομέα της ελιάς τα θέματα αυτά από τους γεωργού μέχρι τη δημόσια διοίκηση, μέχρι τα συνδικάτα ε, και την ίδια την εργοδοσία και θα πρέπει με την ίδια πειθό και την προσπάθεια που έγινε ε, για το χάλιβα και το αλουμίνιο να δοθεί μάχη. Και εντωμεταξύ Μέχρι να συζητηθώ το θέμα των δασμών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβλέψει μέτρα όπως για παράδειγμα αποζημιώσει και βοήθεια για τον τομέα της ελιάς από τη ζημία που προκαλείται και που οι συνέπειες, ε, για άλλη μια φορά επιμένω, ε, πληρώνονται από τους ίδιους τους εργαζομένους. Πρέπει να αναζητηθούν νέες αγορές για αυτή την παραγωγή ποιότητας και να μην ε, ζημιωθούν όπως ζημιώνονται αυτή τη στιγμή η παραγωγή της Σεβίλης. Έχουμε πάρα πολλέ θέσει εργασίας, ακόμα και 2.000 θέσεις μπορούν να χαθούν άμεσα άμεσα ή έμεσα και η ε, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις ε, οι οποίες πλήττονται από τις ε, λύσεις ε, που επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ. Συσκευασία, ο μηχανισμός επεξεργασίας της ελιάς, οι μεταφορείς, ακόμα και οι μηχανικοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις υποδομές και για τους συνεταιρισμούς. Και ολοκληρώνω, εάν δεν επιληθεί αυτό το ζήτημα θα πρέπει να τεθούν επιτάπητος όλες οι διμερείς σχέσεις της χώρας που κυβερνά ο Τραμπ. Μεταξύ αυτών και το θέμα άμυνα. Υπενθυμίζω ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 342 ε, αμερικανικέ εγκαταστάσει, 5 εξ αυτών στην ε, ε, Ισπανία και 2 στην περιοχή τη Ανδαλουσία. Η μία είναι η στρατιωτική βάση του Μωρών και πραγματικά ο οικονομικό μοχλό του είναι ακριβώ αυτέ οι επιτραπέζιε ελιέ τη Σεβίλη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ και τώρα να περάσουμε στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε δύο μέλη της Επιτροπής την κυρία Κοροδήμα και τον κύριο Ε, Έχουμε από τη Γενική Διεύθυνση Τρέι την κυρία Κοροδήμα και μετά ένα εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση Γεωργία. Παρακαλώ, κυρία Κοροδήμα. Κύριε Okay, don't Α, ο κύριο Παβόν πρώτα. Gracias, ε, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Ισμαήλ Σάντσεθ ε, για αυτή την παρουσίαση. Θα μιλήσω αγγλικά τώρα για την παρουσίασή μου για να γίνω κατανοητός γενικότερα για αυτή την ε, αναφορά η οποία διαρκεί 1,5 έτος ήδη την από λίγο καιρό χρησιμοποιού... και πάλι συζητούσαμε τα θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, μπορώ να πω ότι η Κομισιόν συμμερίζεται τις περισσότερες από τις απόψεις σας. Πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι αυτές οι έρευνες γίνονται υπό το πρίσμα της ε, διοίκησης Τραμπ που γενικά έχει θέματα όχι μόνο με εμά αλλά και με άλλε χώρες, άλλους εμπορικού εταίρους. Η διαδικασία της έρευνας, της διερεύνησης δεν ήταν εύκολη. εύκολη. Οι συνάδελφοι στην ε, Γενική Διεύθυνση Trade που έχουν εμπειρία με τέτοιου είδους διερευνήσεις και είπαν ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο τους. Η Αμερικανική διοίκηση ήρθε με τεράστια ποσότητα πληροφοριών και αδιανόητες προθεσμίες. Υπήρξε ένας συντονισμός μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών στην Μαδρίτη και της ε, Κομισιόν αλλά και της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας και των εταιριών. Αλλά παρά τις προσπάθειες αυτές η διοίκηση Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει και να επιβάλλει αυτούς τους δασμούς. Δεν είναι μόνο αυτά που κάναμε στην Κομισιόν, αλλά ε, είχαμε και τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες που έστειλε επίσημες επιστολές στις, στους επικεφαλείς ε, των αντίστοιχων επιτροπών Γεωργίας ε, και Εμπορίου στο κοινοβούλιο τους ε, και τους ζητούσε να σκεφτούν διπλά πριν κάνουν κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, δεν είναι η μόνη που δίνει τέτοιες επιχορηγήσεις στη Γεωργία και οι Ηνωμένε Πολιτείες δίνουν αυτές τις επιχορηγήσεις Green boxes στην Γεωργία. Παρά λοιπόν όλες τις προσπάθειες, ε, τις επιστολές, ε, τις συναντήσεις, ακόμα και ε, η Επιτροπή με εκπρόσωπο τον Επίτροπο Χόγκαν μπόρεσε να συναντηθεί με τους Αμερικανούς. Παρά λοιπόν όλες αυτές τις προσπάθειες, δεν καταφέραμε κάτι και τώρα βλέπουμε στην Εστρεμαδούρα και στην Ανδαλουσία τους Αγρότε να υποφέρουν, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι η κοινή αγροτική πολιτική που υποφέρει, γιατί σύμφωνα με την έρευνα είδαμε ότι κάποιες επιχορηγήσεις όπως το Green, το Skinning, όλα αυτά θα μπορούσαν να επίπτουν να είναι τέλος πάντων ε, λόγος για να επιβληθούν επιπλέον δασμοί. Αυτό είναι λοιπόν ε, top προτεραιότητα και για, για όλες τις σχετικές διευθύνσεις της Κομισιόν. Να πω επιπλέον ότι, όπως αναφέρατε πριν, θα θέλατε να δείτε κάποια αποζημίωση για τον τομέα, αλλά εμείς το εξετάσαμε, ήμασταν ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεχόμαστε ότι υπέφερε ο τομέας και όντως ε, τα στοιχεία που αναφέρατε για την πτώση των εξαγωγών ήταν ξεκάθαρα για μας, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι και ένα από τα πράγματα που κάναμε είναι να, επειδή ξέραμε πως χάσατε την αγορά της μαύρης ελιάς, όχι της πράσινης, στις Ηνωμένες Πολιτείες η Ισπανία, προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε διάφορες ε, δραστηριότητες προώθησης 70 με 80% χρηματοδότηση δόθηκε για εκστρατείες προώθησης που θα διαρκέσουν ένα ή δύο χρόνια και θα τρέξουν σε άλλες αγορές εκτός Ευρώπης ή εντός Ευρώπης, αλλά όχι στις Ηνωμένε Πολιτείε για να μπορέσουν οι αγρότες της Ισπανίας να βρουν νέες αγορές. Σας καλούμε λοιπόν να δείτε τα αναπτυξιακά προγράμματα. Η κοινή αγροτική πολιτική έχει δύο πυλώνες. Πρέπει να κοιτάξετε εκεί και να βρείτε τις ε, επιχορηγήσεις που θα σας βοηθήσουν, τις επιδοτήσεις που θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε. Πρέπει να θυμόμαστε ε, ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να δώσουν 200.000 ευρώ το χρόνο ανά πληττόμενο ε, γεωργό ε, μέσα σε μία περίοδο δύο δημοσιονομικών ετών. Δύο. Τριών, συγγνώμη. Ε, επίσης, ε, δεν υπάρχει ανάγκη να δοθεί άδεια από την Κομισιόν για κάτι τέτοιο. Στο περι... Πολύ αναφέρατε το θέμα της αποζημίωσης ε, στο παρελθόν. Είναι μέσα στα πλαίσια των μέτρων. Ε, όμως ε, το εξετάσαμε και είδαμε ποιες είναι οι πιθανότητες να ληφθούν κάποια μέτρα σε επίπεδο αγοράς για αποζημίωση των γεωργών. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Όταν ξεκινάς τέτοια μέτρα για έναν τομέα, θα πρέπει να ορίσεις πολύ συγκεκριμένα την νομοθεσία, ε, ε, να πρέπει να, είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά στην νομοθεσία. Οι όροι που περιλαμβάνει λοιπόν η νομοθεσία είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν μας επιτρέπουν στην περίπτωση των Ισπανών γεωργών να ξεκινήσουμε τέτοια μέτρα. Δεν μείναμε όμως στο θέμα της πρόθεσης. Περάσαμε και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και θα δώσω το λόγο στη συναδέλφους Έμι και κύριο Λάγκερν για να σας πούνε κάποια πράγματα γι' αυτό. Ναι, ευχαριστώ Σέρτζιο. Όπως εξήγησε ο συνάδελφος από την DG Agri, συνεργαζόμαστε κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας με όλες τις αρχές της Επιτροπής αλλά και τις Ισπανικές αρχές. Δυστυχώς έχουν ήδη επιβληθεί οι δασμοί. Στην απάντησή μας στην αναφορά αναφερθήκαμε το αίτημα για διαβούλευση που είναι το πρώτο στάδιο στην επίλυση διαφορών σε επίπεδο ΠΟΕ Έγινε αυτό, δεν επιλύθηκαν τα ζητήματα και τώρα πήγαμε στο επόμενο βήμα, ένα πάνελ ΠΟΕ που έχει θεσπιστεί, τώρα θα συσταθεί συγκεκριμένα και θα ξεκινήσει σύντομα να λειτουργεί. Το πάνελ αυτό θα εξετάσει το κατά πόσο συμβατά είναι τα μέτρα των ΗΠΑ με τους κανόνες του ΠΟΕ εδώ υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Αυτό που ήδη τόνισε ο αναφέρον και ο συνάδελφος που είναι και συστηματική ανησυχία για μας είναι οι άμεσες ενισχύσεις. Γιατί μπορεί αυτό να εφαρμοστεί και σε άλλα προϊόντα και δεν θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν δασμοί για αυτά γιατί δεν είναι ειδικά. Ένα άλλο θέμα είναι η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, βάσει των οποίων επιβλήθηκαν οι δασμοί, θεωρεί ότι ε, τα ωφέλη περνάνε από αυτούς που καλλιεργούν σε αυτούς που επεξεργάζονται. Επίσης για τον καθορισμό και τον υπολογισμό του ποσοστού υπάρχουν κάποια ζητήματα. Τα κυνηγάμε και αυτά. Είναι όμως μακρά διαδικασία, μπορεί να πάρει ένα χρόνο και για τους Ισπανούς παραγωγούς αλλά και γενικότερα ε, για την ε, κοινή αγροτική πολιτική το θέμα αυτό είναι δύσκολο. Ο κύριος Νάιτζελ Σαλίβα έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου. So here we are witnessing Βλέπουμε λοιπόν μια στρατηγική υπερπροστατευτική και αρκετά ε, επιθετική. Όπως ε, εξήγησα, τα μέτρα είναι δυσανάλογα τελείως. Αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να, ε, να έχουν ως αποτέλεσμα σε ε, μεγάλες απώλειες αρκετών εκατομμυριών ευρώ για τον τομέα. Το χειρότερο όμως είναι ότι, ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα άσχημο ε, προηγούμενο ε, και να ανοίξει το δρόμο για άλλα κράτη-μέλη του ΠΟΕ να ε, αμφισβητήσουν την υπάρχουσα αγροτική πολιτική που θα έχει με τη σειρά του μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να θέσει κίνδυνο το, μοντέλο της, ε, το κρατικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, να, να, να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Γεωργία και να μην περάσουν αυτά τα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε μάλιστα, θα πρέπει να εξετάσουμε όλους τις οδούς ε, ε, Αποζημίωση των αγροτών που έχουν πληγεί από αυτή την στρατηγική. Ευχαριστώ εξ ονόματος του ΕΛΚΟ κύριο Σόιδα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ε, ε, αναφορές τους και συμφωνώ εξ ονόματος του ΕΛΚ πλήρως με τα όσα είπα αναφέρον ότι οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ για τι ε, μαύρε ελές οι οποίε εισάγονται από την Ισπανία αποτελούν πλήγμα για τον κλάδο. Πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για την Ισπανία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα ε, παραγωγό επιτραπέζια ελιά. Έχει το 51% τη παραγωγή παγκοσμίω ε, και η Ανδαλουσία είναι η πρώτη περιφέρεια τη Ισπανία, με περίπου 80% του συνολική παραγωγή. Αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι η Σεβίλη, η Κόρδοβα, η Μάλαγα και το Κάθερες. Και οι απώλειες φτάνουν ε, σε πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ και πιστεύουμε ότι φέτος οι απώλειες θα είναι πολύ περισσότερες διακυβεύονται πάνω από 10.000 ε, άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες εξαρτώνται από αυτές τις εξαγωγές. Και θα θέλαμε εδώ να επισημάνουμε ότι δεν πρόκειται για μία απειλή που αφορά μόνο το συγκεκριμένα τα ε, κλάδο της επιτραπόζιας ελιάς, ούτε καν για αποκλειστική απειλή για την Ισπανία. Αυτοί οι δασμοί της ε, κυβέρνησης των ΗΠΑ θέτουν ένα αμφιβόλο όλο το σύστημα ενισχύσεων της ΚΑΠ το οποίο αναγνωρίζεται ευρύτατα και υποστηρίζεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Γι' αυτό ακριβώ μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα πείραμα το οποίο θα μπορούσε να έχει συνέπειε σε όλη την Ευρώπη. Και ολοκληρώνω λέγοντα ότι θέλουμε με πολύ αποφασιστικό τρόπο να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη και την ε, ε, καταγγελία στον ΠΟΕ, ελπίζοντα ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα όπω μα ανακοινώθηκε, προκειμένου να ε, πάψουν να υπάρχουν οι δασμοί ε, για του οποίου διαμαρτυρόμαστε εδώ σήμερα. Δεύτερον, το ΕΛΚ θεωρεί ότι θα πρέπει να πιοζημιωθούν η παραγωγή του και οι επιχειρήσει του κλάδου τη επιτραπέζια ελιά με έκτακτα μέτρα, λαμβάνοντα υπόψη τα 5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δαπανήθηκαν για ένα σκοπό ο οποίο ε, δεν είναι ε, ευρωπαϊκός και μόνον. Θα πρέπει επίσης να μην ξεχάσουμε ότι δεν θα πρέπει να πληγεί ένας τομέας ε, ο οποίος αποτελεί επίθεση τελικά για όλη την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα έχει το λόγο η κυρία Ροντρίγεθ από το Renew Europe. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ναι, ήθελα να λάβω το λόγο για να υποστηρίξω την πρόταση του αναφερομένου και επίσης ε, τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στην ε, διαμάχη αυτή, αλλά επίσης και να ζητήσω μεγαλύτερη προσπάθεια και μια καλύτερη απάντηση. Ε, όπως μόλις ακούστηκε, η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός επιτραπέζιας ελιάς. Και έχουμε και μια πολύ σημαντική αγορά, Εξαγωγέ προ τι Ηνωμένε Πολιτείε. Η Ανταλουσία παράγει πάνω από το 80% τη Ισπανική παραγωγή και η μαύρη ε, ισπανική ελιά ε, αποτέλεσε στόχο των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Ελήφθησαν αδικαιολόγητα και δυσανάλογα μέτρα τα οποία είναι και ε, σε παραβίαση των κανόνων του ΠΟΕ. Παραβιάζουν τους κανόνες διότι ε, μέχρι σήμερα όπως ε, πολύ σωστά ακούστηκα και από τους δύο εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει περάσει πάνω από 1,5 χρόνος και δεν υπάρχει καμία απόδειξη απολύτως, ούτε επαρκής ούτε ανεπαρκής, ότι η εισαγωγή ε, ισπανικών επιτραπέζιων ελιών έχει επιβαρύνει τον ε, τομέα παραγωγής των ΗΠΑ. Η τιμωρία ουσιαστικά που επιβάλλεται στην Ισπανική Επιτραπέζια Ελιά, ε, τη Μαύρη Ελιά, είναι λόγω πολιτικής απόφασης ε, προστατευτισμού των ΗΠΑ ενισχύσεις τη κοινή γεωργικής πολιτικής και κυρίως οι ενισχύσεις που δίνονται στο συγκεκριμένο κλάδο, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν αποτελούν κίνητρο για την παραγωγή, διότι δεν είναι συγκεκριμένε ενισχύσεις για τον κλάδο, δεν αποτελούν κίνητρο για τις εξαγωγές και δεν σχετίζονται και με την τιμή του προϊόντο Ακριβώ γι' αυτό το λόγο εμπίπτουν στο πράσινο κουτί του ΠΟΕ και επιτρέπονται διότι δεν υπάρχει αντίκτυπος για το διεθνές εμπόριο. Αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Γι' αυτό ακριβώ γνωρίζει και ότι τα συμπεράσματα τη ειδική ομάδα εργασία που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να είναι άλλα ε, παρά το να δηλώσουν σαφέστατα ότι είναι παράνομοι οι δασμοί που επιβάλλονται από τις ΗΠΑ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η συμπεριφορά της ε, αμερικανικής κυβέρνησης ήταν σαφώς να παρακολύσει τη διαδικασία, καταρχάς τις διμερείς διαπραγματεύσεις εντός του ΠΟΕ και ε, δεύτερον της σύστασης αυτής της ομάδας εργασίας, η οποία κατόπιν ετήματος ε, και μετά από τα προσκόμματα που έδωσαν την πρώτη φορά, τελικά συστήθηκε. θα ήθελα να πω όμως ότι ε, και εδώ συμφωνώ και με αυτά τα οποία ακούστηκαν προηγουμένως, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διευκολύνει την ε, ε, απόφαση αυτής της ομάδας εργασίας και πρέπει επίσης να εξετάσει και το θέμα της αποζημίωσης για τις τεράστιες ζημίες που έχουν ήδη υποστεί η παραγωγή και όπως ακούστηκε βρισκόμαστε και ενώπιον μιας προοπτικής διότι έχει χαθεί 1,5 χρόνο δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να αφήσει μόνο του ένα κλάδο, ο οποίο τιμωρείται, λαμβάνοντα υπόψη όλη την κοινή γεωργική πολιτική και τον τομέα των ενισχύσεων, και πρέπει επίση να απαντήσει ε, για τι ζημίε που έχουν ήδη υπάρξει, διότι δεν πρόκειται για το προϊόν αυτό καθεαυτό, πρόκειται για πάρα πολλού παραγωγού, για πάνω από 10.000 θέσει εργασία οι οποίε διακυβεύονται και επομένω πρόκειται για την οικονομία πολλών οικογενειών και για την οικονομία τη υπέρ υπαίθρου πολλών δήμων ε, στους οποίους ε, η παραγωγή και η μεταπίεση της μαύρης ελιάς είναι ε, ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση των οικονομιών τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Αρέγο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρέγο, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ επί τη ευκαιρία θα ήθελα να ζητήσω να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Πιστεύω ότι υπάρχει ε, συνένεση από την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων. Ε, για μέτρα αυτού του ύψους και αυτού του τύπου, το είπε άλλωστε εξαιρετικά και ο αναφέρον, δεν είναι μόνο ε, ο αντίκτυπος που υπάρχει για τις διάφορες περιοχές και τους εργαζομένους, αλλά και για την ανάπτυξη και την ιδιαιτερότητα μιας περιοχής η οποία εξαρτάται οικονομικά από τη συγκεκριμένη παραγωγή και αυτό το προϊόν. Και επίσης να πω ότι δεν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι μεμονωμένο σε τοπικό επίπεδο, αλλά υπάρχουν και άλλοι, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ε, τίθενται εν κινδύνο και όλα όσα έχουν σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο είναι μεγίστη σημασία. Εν τω μεταξύ όμως, μέχρι να επιληθεί, μέχρι να ε, βρεθεί με ποιο τρόπο θα βρεθεί μια λύση σε αυτό το αδιέξοδο και εδώ ε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει κάποιο συμβιβασμό και να υπάρξει παρακολούθηση και να είναι αποτελεσματική η ενίσχυση που θα δοθεί, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και να μην ε, ξεχάσουμε κανένα γεωργό άνδρα και γυναίκα ή συνεταιρισμό που εξαρτάται από τον κλάδο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν βοήθεια, πραγματική βοήθεια και να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ και τώρα η κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναφέροντα, ο οποίος αυτή τη φορά ε, μας φέρνει προς συζήτηση ε, μια κατάσταση, όπως είπαν ε, οι συνάδελφοι, η οποία προέκυψε από τους δασμούς που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε και ψήφισμα, έγιναν πολλά διαβήματα. Εδώ και δύο χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα και εδώ θα ήθελα να προσθέσω, για να μην επαναλάβω πράγματα στα οποία συμφωνούμε όλες οι πολιτικές ομάδες, όλοι όσοι ε, μίλησαν ε, με βρίσκουν σύμφωνοι, επομένω δεν θα επεκταθώ. Ε, θα ήθελα να μιλήσω για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν ετέθη ε, το θέμα των δασμών και επιβλήθηκε προβλήθηκαν αυτοί οι βιασμοί και στο αλουμίνιο και στο χάλιβα δεν επέδειξαν την ίδια ευαισθησία με την ελιά όπως και με το αλουμίνιο και το χάλιβα. Καταλαβαίνω ότι η οικονομική κλίμακα δεν είναι ίδια, αλλά οι ε, συνέπειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες ε, ε, μπορεί να οδηγήσουν και σε ε, κατοπινές συνέπειες, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απειλή ε, για επιβολή νέων δασμών από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να είναι ολέθριες. Ε, ίσως λοιπόν θα πρέπει να καταδείξουμε ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα της Ισπανίας, της Ανδαλουσίας και της Σεβίλης, αλλά είναι ένα πρόβλημα με τις ενισχύσεις ε, της ΚΑΠ. καθυστερήσαμε να το δούμε, αλλά τελικά το διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα αυτό που ισχύει είναι ότι υπάρχουν συνέπειες για τις επιχειρήσεις καταρχάς, εκμεταλλεύσεις οι οποίες πάνω από 50 χρόνια ε, ήταν εγκατεστημένε στι Ηνωμένες Πολιτείες με μεγάλο κύρο γι' αυτό και τιμωρήθηκαν αυτέ οι επιχειρήσεις ε, και υπέδειξαν τρει συγκεκριμένε επιχειρήσεις. Δεν τυχαίο αυτό. Υπήρχε κυριαρχία στην Αμερικανική αγορά ε, και μάλιστα υπάρχουν επενδύσει στο θέμα αυτό για πάνω από 50 χρόνια. Γι' αυτό ακριβώ και έγιναν αντικείμενο στόχο αυτέ οι επιχειρήσει και υπέδειξαν τρει επιχειρήσει. Αυτέ οι τρει επιχειρήσει οι οποίε κυριαρχούσαν στην αγορά με τους δασμούς ε, τελικά εκδιώχθηκαν από την αγορά. Αυτός ήταν ο στόχος ε, των μέτρων Τραμπ. Ε, τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε το θέμα στον ΠΟΕ. Είναι αλήθεια ότι είναι μακροχρόνια διαδικασία. Χαιρόμαστε. Το ζητήσαμε εμεί από πλευρά Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο Εδώ υπάρχει ομοφωνία σε όλε τι πολιτικέ ομάδε και είναι πολύ καλό το γεγονό ότι ε, συνεχίζουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και ε, τα μέτρα είναι ελάχιστα. Ε, οι αποζημιώσει που δίνονται είναι αυτά τα οποία δίνει η Ισπανική κυβέρνηση ή το πρόγραμμα τη ανάπτυξη υπαίθρου, αυτά τα οποία πληρώνουν δηλαδή υπόλοιποι γεωργοί. Θα πρέπει κάπως να καθορίσουμε συγκεκριμένα στήριξη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους οι οποίοι μπορεί να ε, τιμωρηθούν τελικά γιατί η αγορά των ΗΠΑ ήταν η βασική τους αγορά και τελικά η ίδιοι γεωργοί διότι χάνεται ένας μεγάλος συνεταιρισμός με πάνω από 2.000 εταίρους και καταλαβαίνετε ότι οι συνέπειες για την περιοχή είναι ε, καταστροφικές. Ολοκληρώνω λέγοντα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά έκανε κάποια πράγματα. Το Κοινοβούλιο με ομοφωνία των πολιτικών ομάδων βοήθησε πολύ. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω με αυτή την ομοφωνία, να ευχαριστήσω τον αναφέροντα, ο οποίο ε, έθεσε το θέμα επιτάπητο και ε, ζητώ και εγώ να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και ε, να πρέπει να δοθούν ε, ε, βοήθεια είτε από την Ισπανική κυβέρνηση είτε από τους υπόλοιπους γεωργούς. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη βοήθεια για κάτι το οποίο είναι φρικτά άδικο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πριν ολοκληρώσουμε θα ήθελα να δώσω δύο λεπτά το λόγο στον αναφέροντα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ για τη βοήθεια της Επιτροπής σας ε, και για όλες τις παρεμβάσεις ε, και για τα μέλη της Επιτροπής σας και για τους ευρωβουλευτές που έλαβαν το λόγο. Ανεξάρτητα από τα μέτρα αποζημίωση ε, τα οποία δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα είπε ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορέσουν ε, να δοθούν οι αποζημιώσει, ε, βάσει και του γεγονότο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε ότι απογοητεύτηκε από του δασμού που επιβλήθηκαν από τι Ηνωμένε Πολιτείε και φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση υποστήριξη από όλου του Ευρωβουλευτέ που έλαβαν σήμερα το λόγο και που αποδείχθηκε ότι στο θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μια ενιαία φωνή, μιλούν όλοι με μια φωνή, ε, θα ήθελα να ζητήσω αυτή η μία φωνή να μετατραπεί σε δράση. Γι' αυτό λοιπόν κυρία Πρόεδρε σας ζητώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά μέχρι να μάθουμε ε, πώς θα επιληθεί η διαφορά την οποία συζητήσαμε και αναγνωρίζοντας ε, και υποστηρίζοντας τους πάνω από 10.000 εργαζομένους ε, στον τομέα της επιτραπέζιας μαύρης ελιάς στη Σεβίλη. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Σάντσες ε, για την αναφορά σας και για αυτή την παρουσία σας εδώ σήμερα ε, για να μας παρουσιάσετε την αναφορά σας. Μετά από τα όσα ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, από τον αναφέροντα και από τα μέλη ε, ευρωβουλευτές της Επιτροπής, ε, δεδομένης και της ομοφωνίας της Επιτροπής για τη συγκεκριμένη αναφορά, η πρόταση της Προεδρίας είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και επίση θα ήθελα να ευχαριστήσω από πλευρά Επιτροπή Αναφορών ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα έκανε για την ε, προάσπιση του ισπανικού τομέα τη Μαύρη Επιτραπέζια Ελιά, αλλά επίση και τη ε, κοινή αγροτική πολιτική. Γι' αυτό ακριβώ η πρότασή μα είναι να υπάρξει στενή παρακολούθηση τη. Ε, ε, προσφυγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΠΟΕ. Ε, είναι σίγουρο ότι είναι μια ε, αργή διαδικασία, αλλά ζητάμε να μας δώσετε όποια πληροφορία υπάρχει από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επιτροπή Αναφορών για το πώ ε, ε, προχωρά το θέμα τη προσφυγή ενώπιον του ΠΟΕ. Επίση, ε, θα θέλαμε να μα ενημερώσετε και για όλε τι αποφάσει οι οποίες εγκρίθηκαν όσον αφορά τι ενισχύσει, διότι όπω ήδη ακούστηκε στην αναφορά αυτή δεν τίθεται μόνο εν κινδύνο ο ισπανικό κλάδο, αλλά θέτει εν κινδύνο και όλη την κοινή αγροτική πολιτική. Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση τη Προεδρία Επιτροπή τη συγκεκριμένη αναφορά. Ευχαριστώ πολύ και να πω στα όλα τα μέλη της Επιτροπής ότι πρέπει να αποχωρήσω διότι έχω ψηφοφορία. Α, τελείωσε. Οπότε θα παραμείνω με την τελευταία αναφορά στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για την 894 του 2017 από μια Ιταλίδα για την ασύμετρη εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων στη Γερμανία σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονό που αλλοιώνει την κατάσταση τη κοινή αγορά. Η αναφέρουσα δεν είναι παρούσα, μα είπε ότι δεν θα παρευρεθεί στην ε, συνεδρία τη Επιτροπής. Γι' αυτό ακριβώς ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Σαλίμ Μετκούλ, για να μας πει τα της αναφοράς. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η αναφορά έχει να κάνει με τους κανόνες της ε, συνθήκης που αφορούν στις κρατικές ενισχύσεις. Όπως θα γνωρίζει πολύ καλά η Επιτροπή προφανώς, ο γενικός κανόνας υπό τη συνθήκη είναι ότι οι κρατικές ενισχύσεις απαγορεύονται. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις που ορίζονται στη συνθήκη όπου μπορεί να χορηγηθεί κρατική ενίσχυση. Αυτή η αναφορά σχετίζεται με μία από αυτές τις εξαιρέσεις. Είναι το άρθρο 107.2c που αναφέρει ότι μπορεί να δοθεί κρατική ενίσχυση σε περιοχές της Γερμανίας που έχουν πληγεί από την επανένωση της Γερμανίας προκειμένου να ε, υπάρξει μια ε, ανάκαμψη από τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω αυτής της επανένωσης. Ανησυχεί η Κομισιόν διότι μια τέτοια διάταξη μπορεί να οδηγήσει σε μη ισότιμη μεταχείριση συγκεκριμένων κρατών, γιατί κάποια κρατήδια της Γερμανίας ε, μπορεί να λαμβάνουν περισσότερες κρατικές ενισχύσεις από ό,τι είναι δυνατό σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν ε, θεωρεί πως η αναφορά αντικατοπτρίζει μία ανάγνωση της διάταξης που δεν ε, συνάδει με ε, το σκοπό της και τον τρόπο που ερμηνεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέτασε αυτή τη διάταξη πολλές φορές και το, την ερμήνευσε με ένα πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Έχει θέσει δηλαδή όρια στο πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη. Πρώτον, μπορεί να επιτρέψει μια ενίσχυση μόνο όταν είναι τρόπος να υπάρξει αποκατάσταση μειονεκτημάτων που προκύπτουν από την επανένωση ξεκάθαρα. Π.χ. ο σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών της χώρας. Αυτό έχει να κάνει με πράγματα που ίσχυαν το 57. Άρα πρέπει να υπάρχει πολύ συγκεκριμένη σύνδεση με την ε, διάσπαση, ας πούμε, της ε, Γερμανίας. Κάτι άλλο που φαίνεται από την ομολογία είναι ότι σήμερα οι διαφορές ε, σε επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ του δυτικού και του ανατολικού τμήματος της Γερμανίας, μεταξύ δηλαδή των κρατηδίων που ήταν στην παλιά Ανατολική Γερμανία, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, και των κρατηδίων που ήταν στη λαϊκή, στην πρώην Δυτική Γερμανία. Οι διαφορές στην ανάπτυξη λοιπόν δεν είναι βάση για κρατική ενέσχυση υπό αυτή τη διάταξη. Άρα, ο τρόπος που εφαρμόζεται αυτό το άρθρο βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου πρέπει να είναι να υπάρχει άμεση σύνδεση, άμεση συσχέτιση με το κόστος που προκύπτει λόγω της επανένωσης των δύο Γερμανιών. Φαίνεται ότι αυτό του είδους το κόστος δεν ισχύει πλέον, άρα δεν εφαρμόζεται διάταξη. Βέβαια, η επανένωση της Γερμανίας έγινε πριν από 30 χρόνια. Και κατά τη γνώμη μας, θα ήταν δίκαιο να πούμε ότι πλέον δεν έχει πρακτικά κάποια σημασία αυτή η διάταξη και δεν έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις σε κρατικό επίπεδο ε, τα τελευταία χρόνια, ε, τουλάχιστον μετά από την συνθήκη της Λισαβόνας. Κατά την άποψη λοιπόν της Κομισιόν δεν είναι ακριβές να λέμε ότι η διάταξη του 107.2c της συνθήκης θα οδηγεί σε αν, ανισομερή αντιμετώπιση των κρατών μελών και θα θέτει σε κίνδυνο την εσωτερική αγορά. Σήμερα την διάταξη αυτή πρέπει να τη βλέπουμε ως μια ιστορική διάταξη που είχε κάποια λειτουργία σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή αλλά ευτυχώς η ιστορία την έκανε πλέον παροχημένη. Άρα δεν θεωρούμε ότι υπάρχει βάση για αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος που θέλει το λόγο. κύριος Φράουκ este clar că avem de clare atât din partea Curții Europene. Ναι, eh, χρειαζόνται συγκεκριμένες απαντήσεις και έχουμε και συγκεκριμένη απάντηση και από την Κομισιόν και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο αναφέρον μιλάει ε, για έλλειψη υποστήριξης. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να κλείσουμε αυτή την αναφορά εν ώψη των όσων μας είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Εύη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαι διαφορετική άποψη σε σχέση με τον συνάδελφο, γιατί ε, ξεκινώ από μια ουσιαστική πτυχή σε σχέση με τα όσα λέει και ο αναφέρον. Ε, βάσει των επίσημων στοιχείων, των επικαιροποιημένων επίσημων στοιχείων, η περιοχή της Γερμανίας που σήμερα χαίρει κάποιων παρεκκλήσεων για τις κρατικές ενισχύσεις που ακόμα και αν ε, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από ό,τι φαίνεται σήμερα, αλλά επισήμως υπάρχει αυτή η δυνατότητα και προβλέπεται στις συνθήκες, ε, μέχρι σήμερα οικονομικά ε, ευημερούν πολύ περισσότερο από άλλες περιφέρειες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποχρεούνται να σέβονται ε, καθ' ολοκληρίαν ε, την νομοθεσία κρατικών ενισχύσεων. Επομένως, η διάταξη του 107.2 παράγραφος Γ της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που λέει ότι υπάρχουν παρεκκλήσεις οι οποίες αιτιολογούνται από τις ε, οικονομικέ δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η πρώην Ανατολική Γερμανία είναι πλέον αναχρονιστικές. Επομένως, ε, έχουμε φτάσει στα άκρα ε, και θεωρώ ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για να καταργηθούν και προβλέπεται και από τη συνθήκη της Λισαβόνας που το αναφέρει στο σχετικό άρθρο. Εμείς ε, πιστεύουμε όμως ότι όλες οι περιφέρειες θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και εδώ φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να εκφράσουμε πιο αυστηρή άποψη, κάθε άλλο. Και ολοκληρώνω Βάσει των όσων προβλέπονται στις συνθήκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία θα πρέπει να κάνει την πρόταση στο Συμβουλίο ώστε να γίνει η κατάργηση αυτή τη παρέκκληση. Εγώ ελπίζω αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν ώστε να αποφύγουμε ε, στο μέλλον να υπάρχουν ε, προτιμησιακές ε, ε, και καλυμμένες ε, των Γερμανών σε σχέση με του υπόλοιπου πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλό δε μάλλον εάν λάβουμε υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ληκτή στη διαδικασία επιπαραβάση για υπερβολικό χρέος και ζητά μέτρα ε, ε, τεράστιων περικοπών στα κράτη-μέλη. Ποτέ όμως δεν παρενέβη για να επιβάλλει κυρώσεις στη Γερμανία που εδώ και 7 χρόνια δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες ε, μακροοικονομικές ανισορροπίες με τα εμπορικά πλεονάσματα τα οποία είναι πολύ πάνω από το προβλεπόμενο ποσοστό του ΑΕΠ της βάση των κανόνων. Είναι η αλήθεια ότι από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή η συνθήκη τη Λισαβόνα ε, δεν υπήρξε καμία απόφαση για θέματα κρατικών ενισχύσεων βάσει του σχετικού άρθρου. Γι' αυτό ακριβώ ε, θα πρέπει να προτείνουμε την κατάργησή του σήμερα, ε, διότι αυτό δεν θα υπάρξει καμία συγκεκριμένη, δεν θα οδηγήσει καμία συγκεκριμένη συνέπεια. σα ίσα θα βρει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνη, γιατί θα υπάρξει αξιοπιστία και θα θεωρηθεί ότι φερόμαστε ισότιμα σε όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Ζήτω λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά η κυρία Σντάνοκα. Και εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τέτοια ίδια επιχειρήματα με την κυρία Εύη. Ναι, η ιστορία είναι ιστορία και είναι περίπλοκη, όμως ήταν περίπλοκη και για όλη την Ευρώπη. Είναι πραγματικά λοιπόν αυτά τα επιχειρήματα για τις παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, οπότε επαναλαμβάνω τα ίδια επιχειρήματα και προτείνω να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αυτή την ε, επαυτή της αναφοράς και να μην την κλείσουμε τώρα. Κυρία Κέρντον. Ναι, και εγώ συμφωνώ με τη συνάδελφο από το ΕΛΚ. Η απάντηση της Επιτροπής ήταν ξεκάθαρη. Διάφορα ζητήματα εμπλέκονται και αναμειγνύονται στα συζητήσεις για τις κρατικές ενισχύσεις. Υπάρχουν διάφορα θέματα που προκύπτουν ε, όταν συζητάμε τέτοιες υποθέσεις. Ε, υπάρχουν ξεκάθαροι καλώνες και υπάρχει και μια πολιτική και εθνική διάσταση που εμπλέκεται στη συζήτηση. Ήταν ξεκάθαρη λοιπόν η απάντηση της Επιτροπής και προτείνω να κλείσει η αναφορά. Ευχαριστώ πολύ μετά από τα όσα ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, έχοντας διαβάσει και την αναφορά του αναφέροντος και ακούγοντας και τα μέλη, η πρόταση της Προεδρίας είναι να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώθηκε εξέταση αυτής της αναφοράς και να κλείσει, διότι τα μέτρα ε, αφορούν ε, το δίκαιο και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επομένως, με αυτό ολοκληρώνεται και σήμερα το απόγευμα η συνεδρία τη Επιτροπής Αναφορών. Αύριο το πρωί στις 9 η ώρα θα συνεχίσουμε τη συνεδρία τη Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.